Allora, la seduta è aperta. Άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη προβλέπει δηλώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Επιτροπή σχετικά με τα συμπεράσματα τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 17η και 18η Οκτωβρίου. Προτού ξεκινήσει όμω η συζήτηση, πρέπει να σα πω ότι προκειμένου να πάρετε τον λόγο με τη διαδικασία Catch the Eye, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλέν κάρτα είτε με την συμβατική διαδικασία ή με το νέο σύστημα το οποίο σας επιτρέπει να εγγραφείτε στον κατάλογο μιλητών ηλεκτρονικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γι' αυτό την κάρτα ψηφοφορίας και σας προτρέπω να το κάνετε αυτό το συντομότερο δυνατό και να μην περιμένετε αναγκαστικά το τέλος της συνεδρίασης. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Τούσκ. Ντόναλτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντάβιντ. Πρόεδρε σας όλοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την τελευταία μου έκθεση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ας επικεντρωθούμε σε τρία ζητήματα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε τη μονομερή στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία. Κανείς πραγματικά δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία. Θα πρέπει με μόνιμο τρόπο να σταματήσει η Τουρκία την στρατοτική της δράση σεβόμενη το διεθνές δίκαιο. γιατί στη διαφορετική περίπτωση έχουμε μια παράδεκτη ανθρώπινη οδύνη, νίκη της Δάες, καθώς επίσης και σημαντικότατες απειλές όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης τόνισε την πλήρη ελεγγύη του με την Κύπρο που αντιμετωπίζει τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας. Όσον αφορά τώρα το Brexit, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μέσω της διαπραγματικής ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, βάσει της συμφωνίας που εγκρίναμε με την προηγούμενη κυβέρνηση, η αλλαγές που έχουν να κάνουν με το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που ονομαζόταν στο παρελθόν backstop έχει τώρα τροποποιηθεί ο Πρωθυπουργό Τζόνσον αποφάσισε ότι θα μπορούσαν να γίνονται τελειωνιακοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου τη Βόρεια Ιρλανδία, προκειμένου να μην έχουμε τέτοιου ελέγχου μεταξύ Βορείου Ιρλανδία και Ιρλανδία. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και την ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά. Η αναθωρημένη λοιπόν αυτή συμφωνία ήταν αποδεκτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρώτον είχε την υποστήριξη τη Ιρλανδία, δεύτερον είχε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά αυτόν τον τρόπο όλοι οι διαπραγματευτικοί μας στόχοι πληρούνταν και τρίτον διότι αποφεύγεται κατά αυτόν τον τρόπο μια μη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευρά του Συμβουλίου ολοκληρώσαμε τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν και το νομικό πλέον κείμενο έχει έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα που πρέπει να δραματίσει ένα καθοριστικότατο ρόλο η κατάσταση είναι αρκετά πολύπλοκη, ιδίω μετά τι εξελίξει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για μια περαιτέρω επέκταση τη όλη διαδικασία. Εγώ αυτή τη στιγμή έρχομαι σε επαφή με του αρχικού κρατών κυβερνήσεων για να δούμε πώ θα αντιδράσουμε και θα λάβουμε μια απόφαση τι επόμενε ημέρε. Είναι σαφέ ότι τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από αυτό το οποίο θα αποφασίσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, δεν θα αποφασίσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Ένα πράγμα όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφές, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό Τζόνσον ε, το Σάββατο, ένα Brexit χωρίς συμφωνία δεν θα αποτελέσει ποτέ δική μας απόφαση. Τέλος, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάνανε μια πολύ δύσκολη συζήτηση όσον αφορά τη διεύρυνση μετά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών ήθελα να ξεκινήσουν ταξιακές διαπραγματεύσει με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ομοφωνία την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά την άποψή μου αυτό συνιστά σφάλμα και το έχω πει αυτό στους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων και μάλιστα με έναν τρόπο ακόμα πιο άμεσο και ρητό. Ελπίζω απλώς τώρα ότι οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων θα καταλήξουν στα σωστά συμπεράσματα όταν συζητήσουν την διαδικασία προσχώρηση πριν την διάσκεψη του Ζάγκρεπ το Μάιο του 2020. Μαζί με την εκλεγήσα πρόεδρε Φόντερ Λέινεν συζητήσαμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη στρατηγική μας ατζέντα, το στρατηγικό θεματολόγιο, το μελλοντικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και τι επερχόμενε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική, δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, όχι μόνο για τον οικονομικό μα τομέα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό για να βελτιώσουμε παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, καθότι είναι η τελευταία μου αγόρευση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία και του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη μου ευγνωμοσύνη προς αυτόν και την εργασία που έχει επιτελέσει. Διανύσαμε πέντε δύσκολα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο καταφέραμε να συνεργαστούμε πάντα καλή την πίστη. Ο διαφορετικό ρόλο που είχαμε και πολλέ φορέ οι διαφορετικέ μα προοπτικέ οδηγούσαν και σε πολιτικέ διαφωνίε. Αυτό που μπορώ να πω όμω, χωρί κανένα ενδιασμό, είναι ότι ο Ζαν Κλοντ ήταν πάντα απόλυτα προσιλωμένο στην Ευρώπη και εξυπηρέτησε πολύ καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πραγματική μου τιμή που μπορώ να σε αποκαλώ φίλο μου. Σε ευχαριστώ πολύ Ζαν Κλοντ. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα πέντε χρόνια πολύ καλή συνεργασίας. Δεν σημαίνει ότι πάντα συμφωνούσαμε. Το αντίθετο μάλλον συνέβαινε. Πάντως πάντα σας σεβόμουν γνωρίζοντας ότι μοιραζόμαστε ένα κοινό στόχο να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή μας Ένωση και τον Ευρωπαϊκό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Τούσκα. Τώρα το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζαν Jean-Claude Juncker. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συνάδελφοι. Ήταν συγκινητική η προηγούμενη εβδομάδα στην, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο παρέστην μαζί με τον Ντόναλτ, το φίλο μου. Συζητήσαμε, ε, συμμετείχα σε 147 συμβούλια στην καριέρα μου. Ίσως και 148, δεν είμαι σίγουρος. Και σήμερα είναι η εκατοστή πεντηκοστή φορά που εμφανίζομαι εδώ ενώπιον της Ολομέλειας. Εδώ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις συμπεριλαμβανόταν και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. θα μπορούσαμε να έχουμε αφιερώσει το χρόνο μας σε άλλα θέματα που θα βελτίωναν την ε, ζωή των πολιτών μας. Ε, η Κομισιόν όμως ε, ακούραστα διαπραγματεύθηκε μια συμφωνία απαχώρησης για το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να σεβαστούμε την απόφαση του Βρετανικού λαού. Τώρα έχουμε μια τέτοια συμφωνία που και πάλι δημιουργεί μια νομική ασφάλεια για μια εφτακτή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άκουσα τον Μπόρις Τζόνσον όπως άκουσα και την προηγούμενη Πρωθυπουργό την κυρία Μέη. Ο κύριος διαπραγματευτής μας, ο κύριος Μπαρνιέ, εργάστηκε επί 24 ώρου βάσεως και απέδειξε την αποφασιστικότητά του και τη δημιουργικότητά του. Η συμφωνία αυτή καλύπτει τα αιτήματα, όλα τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Λυπούμαστε για την αποφάση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορούμε να εκταχτούμε στον καθρέφτη και να είμαστε βέβαιοι ότι κάναμε οτιδήποτε είναι δυνατόν έτσι ώστε αυτή η αποχώρηση να είναι εφτακτή. Και με το ίδιο πνεύμα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως από το τι θα συμβεί από την άλλη μεριά της μάχης. Τώρα παρακολουθούμε την κατάσταση του Westminster πολύ στενά. Δεν θα μπορούσαμε όμως ποτέ να φανταστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικυρώσει αυτή τη συμφωνία πριν το Westminster την έχει επικυρώσει το ίδιο. Δηλαδή πρώτα το Λονδίνο και μετά εμείς. Ε, κύριε Πρόεδρε, ασχοληθήκαμε επίσης με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα ήθελα να φερθώ στα πρακτικά και να πω ότι έχω την ε, γνώμη ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Δεν θα πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Αλλιώς θα περιέλθουμε σε ένα οικονομικό διέξοδο κατά τα δύο πρώτα χρόνια του, πολιτούς, του δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, θα πρέπει οι χώρες μέλη ε, και άλλοι μας εταίροι να γνωρίζουν πιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ισχύει. Για παράδειγμα, οι φοιτητέ του Εράσμους και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοήσουμε αυτούς τους σημαντικούς εταίρους όσον αφορά την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, μόνο και μόνο επειδή μας είναι να πετύχουμε μια συμφωνία. Ε, και θα ήθελα να πω ότι ο, ο προταθής από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν αποτελεί ένα μίνιμουμ. Ε, και οι προτάσεις οι οποίες βρίσκονται τώρα στο τραπέζι της Φιλανδικής Προεδρίας ε, δεν είναι ε, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Δεν είναι δυνατόν να πρικοδοτήσουμε την Ευρώπη με το 1% του ΑΕΠ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κύριε Πρόεδρε, ε, αναφερθήκαμε για την, ε, στη διεύρυνση. Πραγματικά είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος για τη μη λήψη απόφασης στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία είχαν ε, ε, το δικαίωμα να προσδοκούν ότι θα υπάρξει μια έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για βαρύ σφάλμα να μην έχουν ξεκινήσει, να μην έχουν ανοίξει οι διαπραγματεύσεις με αυτές τις δύο χώρες. Πραγματικά πρόκειται για βαρύ σφάλμα γιατί πλήττει δύο χώρες ε, και κατ' ουσία ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει την εντύπωση ότι δίνει ε, υποσχέσεις τις οποίες ε, δεν εκπληρώνει. Και στην περίπτωση αυτή και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Γιούγκερ. Ας ακούσουμε τώρα του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Βέμπερ. Äh, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ντόναλτ Τούσκ για την πενταετή του θητεία, για το έργο που επετέλεσε όσον αφορά τον κοινό ευρωπαϊκό οίκο και πραγματικά πρόσθεσε να εξασφαλίσει μια συνοχή στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σημείωσε πολλά βήματα πρόοδου. Επεσήμανε ότι όλοι ε, τα σώματα υπέρ τη κοινή ιδέα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εντό αυτού του σώματο είναι πιο εύκολο να υπερασπιστούμε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή ιδέα από ότι στο δικό σου ευρωπαϊκό, στο επίπεδο του δικού σου ευρωπαϊκού ευχαριστώ και εκ μέρου του ΕΛΚ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ε, δυστυχώ δεν μπόρεσε να λάβει την απόφαση σχέση με την Τουρκία. Ε, πρόκειται για μια παράνομη, υπό την έννοια του διεθνού δικαίου, εισβολή ε, στα, στο έδαφο τη Συρία θανατώθηκαν πάρα πολλοί ε, Κούρδοι μαχητές ε, και είναι πάρα πολύ κρίμα το ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Έχουμε τις παράνομες γεωτρήσεις στο Αιγαίο, έχουμε καταστολή της ελευθερίας του τύπου, έχουμε την παράνομη εισβολή στην Τουρκία, το προσφυγικό. Πού βρίσκεται εδώ ξεκάθαρο, ε, ε, η ξεκάθαρη χειρονομία εκ μέρου της Ευρώπης. Θα πρέπει να το καταγγείλουμε ε, ρητά. Γιατί πραγματικά ε, λέμε ότι όλα αυτά μας αφορούν, αλλά αυτό δεν αρκεί και έχουμε την άποψη στο βαθμό που η Τουρκία φέρεται τόσο επιθετικά θα πρέπει να συζητήσουμε και για οικονομικές συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμεθα η Τουρκία να επωφελείται από την Τελωνική Ένωση και την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και από την άλλη να δείχνει τόσο επιθετική συμπεριφορά. Δεύτερον, το δεύτερο το οποίο μας αφορά είναι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, οικονομικά θέματα. Η πρόταση της Φιλανδίας συνιστά μια πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Jean-Claude Juncker είπε ότι δεν καλύπτει για την επιτυχή ανταπόκριση σε σημαντικά ευρωπαϊκά προβλήματα. Και το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να ρισκάρει ε, τελικά να αποτύχουν ε, οι προτάσεις που υποβάλλει λόγω ακριβώς της αντίστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει για να ανταποξέλθουμε στα νέα θέματα να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους ε, πόρους. Και ο προϋπολογισμός ε, είναι ένα προσχέδιο, δεν είναι να υπάρξουν τέτοιε περικοπές ε, σε προγράμματα ε, μείζωνος σημασία όπως είναι το Εράσμος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε διαπράξει το ιστορικό σφάλμα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Η Βόρεια Μακεδονία και η Ελβανία στερούνται από την προοπτική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ενώπιον του ερωτήματος κατά πόσο θα πρέπει να εξαγάγουμε σταθερότητα στα Βαλκάνια ή να εισαγάγουμε μια αστάθεια από τη Βαλκανική. Και στο μέτρο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια βαριά αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συνοβουλίου σε σχέση με αυτό το ζήτημα μίσων ιστορική σημασία. Η Βόρεια Μακεδονία χρειάστηκε να αλλάξει την ονομασία τη χώρα τη προκειμένου να έχει μια προοπτική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέβαλαν προσπάθεια, εμόχθησαν και τώρα του κλείνουμε την πόρτα. Πρόκειται για μια βαριά απώλεια τη αξιοπιστία μα ε, και για την οποία θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι επικεφαλεί των κυβερνήσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε πολύ, είμαι πολύ υπέρ του να εξετάσουμε τις ε, δομές μας. Ε, εφόσον ε, βεβαίως δεν τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας. Είχαμε προειδοποιήσει τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Όχι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια πτυχή που αφορά την πολιτική του κόμματό μας. Το ΕΛΚ υπήρξε συσπηρωσμένο όσον αφορά την προοπτική προσχώρηση τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν ε, δύο εκπρόσωποι του Ρινιού, ε, οι οποίοι ε, τελικά στέρισαν αυτή την προοπτική στις χώρες αυτές. Ο ένας από τους δύο ήταν ο Μακρόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όσον αφορά το Brexit, ας ε, περιμένουμε πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ, τσάι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο να μένουν σε εξελίξει στη Βρετανία. Εγώ μίλησα από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένα συμβιβασμός. Ο Μισελ και οι διαπραγματευτέ στο Λονδίνο ε, και ο Τζόνσον βρήκαν ένα συμβιβασμό να μην υπάρξουν σκληρά σύνορα, όχι backstop. Τώρα έχουμε τη διαδικασία στο επίπεδο του, της Βουλής των Κοινοτήτων και της βουλή των Λόρδων και τελικά θα δούμε, αυτή, ε, θα δούμε την έκβαση κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές οι τροποποιήσεις ή όχι. Και για μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα έλεγα ότι έχουμε το ίδιο δικαίωμα να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση του κειμένου το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ανάγκη να επισπεύσουμε τις εξελίξεις, να βιαστούμε. Έχουμε το ίδιο δικαίωμα να το συζητήσουμε στο επίπεδο της ΑΦΚΟ και στο επίπεδο της ε, Ολομέλειας και των πολιτικών ομάδων Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το τελευταίο θεσμικό όργανο το οποίο καλείται να, λάβει την, να, κάνει, να προωθήσει τελική αξιολόγηση όχι μόνο τεχνικής φύσεως αλλά και πολιτική όσον αφορά την συμφωνία. Αλλά οι τελευταίες μέρες θα έδωσαν δυνατότητα εν τέλει να διαχειριστούμε μια σωστή εξέλιξη, ε, μια θετική εξέλιξη όσον αφορά το Brexit. Και υπάρχει μια ευκαιρία τώρα να υπάρξει, να ορσικοποιηθεί η φιλία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέμπερ. Τώρα η κυρία Γκαρσία Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Τούσκ. Και εγώ εποφελούμε προκειμένου να εκφράσω την αναγνώρισή μου προς το πρόσωπό σας ε, και τη δική μου και της ομάδας μου ασφαλώς. Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε σε σύγκρουση με το Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια ε, και σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές ε, κάνατε προκειμένου να εργαζόμαστε για κοινού στόχους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το τελευταίο ε, δεδομένης της επικαιρότητα. Πρώτον το Brexit, δεύτερον η αρχή μιας νέας κοινοβουλευτική ε, περίοδου για την οποία ακόμα δεν έχουμε προπολογισμό. Το Brexit είναι μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία για όλους. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, πάντοτε έλεγαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέλαμε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη διαδικασία κάθε βήμα είναι σημαντικό. Το ίδιο ήταν και το βήμα που έκανε το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό το Σάββατο ε, που ε, ε, ψήφισε μια τροπολογία που έχει ως στόχο να αποφύγει την άτακτη έξοδο. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι το Βρετανικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Μόνο τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες και θα πράξει ανάλογα. Θέλω να ευχαριστήσω τις προσπάθειες του τον Μισελ Μπαρνιέ για τις προσπάθειές του ε, που έκανε να μας κρατήσει ενωμένου. Ε, μόνο ενωμένοι είμαστε δυνατοί. Το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο ε, έδειξε ενότητα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και την ίδια ενότητα θα πρέπει να δείξουμε εν ώψη των επόμενων πέντε ετών. Αν θέλουμε να είμαστε πιστικοί θα πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Στις τελευταίες εκλογές ε, το εκλογικό σώμα μας ζήτησε μια καινούργια Ευρώπη, πιο οικολογική, πιο αποφασιστική σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, ε, με περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα και ισότητα και πιο διαφανή στη λήψη των αποφάσεων. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δείξει περισσότερη ηγετική στάση, ανάλογη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Την Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζήτησε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 να είναι κλιματικά ουδέτερη. Ε, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων θα πρέπει να κάνουν τα αντίστοιχα βήματα. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, κατάφεραν η νέα πράσινη συμφωνία να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της νέας κομισιόν. Αλλά αυτό θα επιτύχει μόνο αν έχουμε και τα κατάλληλα κονδύλια, επαρκή κονδύλια δεν είναι δυνατόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογένειε να πληρώσουν το λογαριασμό της κλιματικής μετάβασης. Θα χρειαστούμε ένα προπολογισμό που θα χρηματοδοτήσει δίκαια αυτή τη μετάβαση. Αυτό μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνο μέσω ενός φιλόδοξου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Το Κοινοβούλιο έχει τις, προτεραιότητε τις ε, του, τις έχει καθορίσει. Τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο. Η στάση μας είναι πάγια. Θα στηρίξουμε ένα προπολογισμό μόνο αν έχει νέου ίδιου πόρου που θα αντικατοπτρίζουν τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε καινούρια εργαλεία για τη χρηματοδότηση πολιτικών που είναι απαραίτητε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεωργία, συνοχή, αλληλεία θα πρέπει να έχουμε επαρκής ε, επαρκή χρηματοδότηση για την ε, άμυνα, την ε, μετανάστευση και να αντιμετωπίσουμε και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες μας. Ως προτεραιότητες της, πρώτης, της επόμενης ε, ε, κομισιόν έχουμε, μια, ε, έχουμε κονδύλια για την εγγύηση για τους νέους, κονδύλια για τα φτωχά παιδιά, κονδύλια για τους ανέργους και για την κοινωνική ασφάλιση. Το σημαντικό είναι η, η Ευρώπη να αναπτυχθεί. Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από το 1,3% του ΑΕΠ ως προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αναλάβει τι ευθύνε τη. Επίσης χάνουμε πιστικότητα όταν χάνουμε αξιοπιστία, όταν δίνουμε υποσχέσεις στους γειτονές μας και μετά τους κρεμάμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ασφαλώς και έχουν πολλά να κάνουν αυτές οι χώρες και οι διαπραγματεύσεις είναι μακρύς δρόμος. Όμως θα πρέπει να αποτελέσουν και ένα σωσίβιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ολοκληρώσουμε την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί αυτό θα βοηθήσει και την σταθερότητα τη περιοχή, αλλά και στην σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση στο διεθνέ πεδίο θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Στηρίζουμε την καταδίκη της Τουρκίας για την στρατιωτική της επέμβαση, παρόλο ότι λυπούμαστε που δεν ελήφθησαν άλλα μέτρα. Και θα ήθελα επίσης να δώσω ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο δεν θα επιτρέψουμε η Τουρκία να συνεχίσει τις παράνομες γεωτρήσεις της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ακαιρεότητα της Κύπρου. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και δέσμευση για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο θα κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος Τσόλος τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, αγαπητέ Ντόναλτ, φτάνει στο τέλος της θητείας σου. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ μαζί σου και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στα πλαίσια του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά βλέπω ότι συμβάλλεις πάρα πολύ επικοδομητικά στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενότητα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά για τα όσα έκανε ε, για την Ευρώπη. Όσον αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Brexit, αρχίζουμε και συνηθίζουμε σιγά σιγά την κατάσταση αυτή. Θεωρούσαμε ότι βλέπαμε φω στο βάθο του τούνελ και τώρα βλέπουμε ότι οι Βρετανοί συνάδελφοι έχουν ιδιαίτερη φαντασία και καταφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο να επιτείνουν συνεχώ την όλη διαδικασία αποχώρηση χωρί να λαμβάνουν τελική απόφαση. Οι φίλοι μας από τη Βρετανία πάντα επέκριναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας ότι είχαν πάντα μια ιδιαίτερα θεσμική δημιουργική στάση. Μα ακριβώ το ίδιο τώρα κάνουν και αυτοί. Τόσο το καλύτερο βέβαια αν η παράταση αυτή είναι για ένα καλό λόγο. Ωστόσο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς ε, χαιρόμαστε γιατί έχουμε πλέον μία συμφωνία αποχώρησης και για να ευχαριστήσω για αυτήν τον Μισελ Μπαρνιέ και όλη την ομάδα του. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να έχουμε αποχώρηση του Μένου Βασιλείου συνοδευόμενη από συμφωνία. Περιμένουμε τώρα η Βουλή των Κοινοτήτων, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, να ολοκληρώσει την εργασία του. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να λάβουμε καμία απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού ληφθεί μια τελική απόφαση και μία επικύρωση της απόφασης αυτής από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά όπως είπε και ο Μάνφρεντ πριν από λίγο, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ασκηθεί πίεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτελέσει το δικό του έργο και σίγουρα δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία τα οποία έθιξε το Συμβούλιο, να αναφερθώ σε δύο ζητήματα, στον προπολογισμό και στη διεύρυνση. Όσον αφορά τον προπολογισμό, η δική μα πολιτική ομάδα συμμετείχε στην σύνταξη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει λοιπόν την ευθύνη του αυτή, όχι μόνο ζητώντα έναν ισχυρό προπολογισμό, αλλά ζητώντα επίση να μην δημιουργήσουμε μια Ευρώπη μόνο βάσει αριθμητικών δεδομένων, αλλά βάσει συγκεκριμένη φιλοδοξία. Ο κοινοτικό προπολογισμό δεν μπορεί απλώ να είναι μια άθρηση των συνεισφορών των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εργαστούμε περισσότερο, να καταφέρουμε να έχουμε δικού μα ίδιου πόρου και να καταφέρουμε να εκπονήσουμε τελικά ένα προπολογισμό ο οποίο να είναι καθαρά ευρωπαϊκό όσον αφορά τη διεύρυνση ως ε, Ρουμάνος υπήκος προερχόμενος από μια χώρα η οποία υποφελήθηκε ιδιαίτερα από τη διαδικασία της διεύρυνσης είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η διαδικασία της διεύρυνσης θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη αν δεν είμαστε ανοιχτοί προς τους ε, γείτονές μας και αν δεν ε, είμαστε ανοιχτοί προ ε, τι χώρε εκείνε που πιστεύουν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλέ φορέ περισσότερο από τα υφιστάμενα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόρτε λοιπόν τη Ένωση πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ και η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσει μια πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη δημοκρατικών προσπαθειών. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τις χώρες αυτές να κάνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς να τους δίνουμε μια συγκεκριμένη φιλοδοξία και μια ξεκάθαρη ιδέα ευρωπαϊκής προοπτικής. Καταλαβαίνω βέβαια τις ανησυχίες που εκφράσαν ορισμένες χώρες, καθώς επίσης και το ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε του ευρωπαϊκού θεσμού και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε την επόμενη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Δεν σημαίνει όμω ότι αυτό θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία διεύρυνση. Οι πρώτε λοιπόν τη Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνουν ορθάνικτε. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. Ο πρόεδρο Λάμπερτ τώρα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πάλι έχω την αίσθηση ότι έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό. Έχουμε ένα déjà vu, όπως είπαν και οι Βρετανοί, για να περιγράψουν την κατάσταση αυτή. Τα έχουμε βιώσει όλα αυτά. Τον Νοέμβριο του 2018 είχαμε τότε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο χαιρέτησε θριαμβευτικά μια συμφωνία με την τότε Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είδαμε όμω τι δεν μπόρεσε τελικά να κάνει το Βρετανικό Κοινοβούλιο με τη συμφωνία αυτή. Άρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Είδαμε διαφορετικέ εκδοχέ τη συμφωνία αυτή και τώρα όλα βρίσκονται στα χέρια τελικά τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι το Βρετανικό Κοινοβούλιο αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, είτε θα επικυρώσει, και το τονίζω αυτό, είτε θα επικυρώσει, όχι απλώς να πει γενικά και άρρωστα τη συμφωνία, είτε θα επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία αυτή και θα επιτρέψει το Κοινοβούλιο να κάνει την εργασία του ή διαφορετικά θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το Συμβούλιο να επιτρέψει και στο δικό μας το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία εξέτασης και επικύρωσης. Ξέρω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σέβονται πάρα πολύ το Κοινοβούλιο μας, μολονότι Πολλέ φορέ έχουμε κάποιε διαφωνίε, υπάρχει ένα πνεύμα αμοιβαία εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, ενδεχομένω το Βρετανικό Κοινοβούλιο να απορρίψει, να μην δεχθεί τελικά να επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή θα πω το εξή. Αν δεν μπορείτε, δεν θέλετε να επικυρώσετε τη συμφωνία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει πραγματικά να έχετε τα κότσια να θέσετε την, την μη συμφωνία αυτή ή ακόμα και την προηγούμενη συμφωνία που αντιπραγματευτήκαμε με την Τερέζα Μέη σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, να αποφανθεί δηλαδή εκ νέου ο Βρετανικό λαό. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε μια απόφαση. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια σαφή βρετανική επιλογή την οποία θα σεβαστούμε και θα τηρήσουμε. Εμεί δίνουμε μάχη για να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν η πλειοψηφία αποδεχθεί τη συμφωνία, τότε εμεί θα τηρήσουμε προφανώς, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή. Να πω και κάποια πράγματα τώρα όσον αφορά τη διεύρυνση. Για μας είναι σαφέστατο ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ευρωπαϊκή προοπτική και πρέπει να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι προ το συμφέρον κανενό, ούτε των πολιτών των χωρών αυτών, ούτε των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αφήσουμε τις χώρες αυτές σε αυτό το καθεστώς εκκρεμότητος. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κατά αυτόν τον τρόπο οι χώρες αυτές θα παρεκκλίνουν από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση τώρα που έλαβε το Συμβούλιο ως προς διαδικασία διεύρυνσης και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα κύριοι Τούσκα και Γιούνκερ, η απόρριψη αυτή ουσιαστικά της ε, ευρωπαϊκής ε, προοπτικής ουσιαστικά αποτελεί ένα σφάλμα, ένα σοβαρό σφάλμα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο καταλαβαίνω ότι χρειαζόταν βέβαια ομοφωνία και συντοπίω ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών του Συμβουλίου ήθελε να προχωρήσει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά το είπε πολύ σωστά ο Μάνφρετ Βέμπερ. Είναι δύο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έλαβαν τελικά την απόφαση να μπλοκάρουν την όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή αναφερόμασταν απλώ στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειτο για ολοκλήρωση και επίσημη προσχώρηση των κρατών μελών αυτών, των κρατών με αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η όλη διαδικασία τη διεύρυνση ξέρετε ότι είναι μια πολύχρονη διαδικασία και απαιτεί πολλά διαφορετικά στάδια. Όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν εκλέγει στη θέση του Προέδρου της ε, Γαλλικής Δημοκρατίας. Χαιρετήθηκε από πάρα πολλούς ως μέγας ε, φιλοευρωπαίος ηγέτης. Ενδεχομένως να μην είναι τελικά τόσο ευρωπαίος ηγέτης ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο κύριος Μπέ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τουρκία ε, το μεγαλύτερο μέρος της ε, συζήτησης του Συμβουλίου εδώ και 45 χρόνια ε, έχει υπό την κατοχή τη, ένα τμήμα τη Κύπρου μια χώρα μέλος την οποία, ε, η οποία δέχεται σφοδρή επίθεση εκ μέρους της Τουρκίας η οποία τώρα θέλει να προβεί σε παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου. Η η Τουρκία παραβίασε το διεθνές ε, δίκαιο επεμβαίνοντας στη βορειοανατολική Συρία και αυτή η δραστηριότητα ενίσχυσε ε, τους διχαντιστές στην Αρνόσα ή το ε, Νταέσο. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 5,6 δις για το προσφυγικό ε, παρόλο που η Τουρκία τελικά πολλαπλασιάζει τις ε, απειλές της, εκβιάζοντας τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και απειλώντας να ανοίξει τις πύλες τους πρόσφυγες. Δώσαμε λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα και σήμερα παρόλο αντί να ε, ανασταλεί η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας είναι απολύτως αναγκαίο να τερματιστεί αυτή η προοπτική γιατί η Τουρκία ε, λόγω του πολιτισμού της και της ε, στάσης της τελικά είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση στο Συμβούλιο αναφέρθηκε επίσης στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και έγινε ε, λόγος ε, για τη φορολογία στον άνθρακα, στο πλαστικό, σαν μοναδική λύση. Ε, υπάρχουν πάντα τα ίδια προσχήματα τα οποία εφαρμόζονται, το, ε, κυρίως το οικολογικό πρόσχημα. Ωστόσο, τι θα μπορούσε να γίνει ε, θα μπορούσαν να πολλαπλαστούν οι συμφωνίες ελεύθερων ε, ανταλλαγών με χώρες οι οποίες δεν ε, δέχονται να σεβαστούν τις προδιαγραφές και με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και πλήττεται η αγοραστική δύναμη των συμπατριωτών μα. Όσον αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε κανεί να συνοψίσει τα πράγματα ω εξή. Να δίνουμε όλο και περισσότερα για να έχουμε όλο και λιγότερα. Η Γαλλία έδωσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια ε, και σαν αποτέλεσμα ε, είχαμε μια πλήρη αποδυνάμωση της γεωργίας. Ε, κάθε δύο μέρες αυτοκτονεί ένας Γάλλος ε, καλλιεργητής, αγρότης. Θα πρέπει να υπάρξουν προστατευτικά μέτρα, είναι αναγκαίο αυτό, αντί να πηγαίνουμε όλο και πιο πέρα στην παγκοσμιοποίηση των ελεύθερων ανταλλαγών. Ο κ. Φανόρντεν, παρακαλώ. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ευελιξία και καλοπιστία σε ό,τι αφορά τον, τον Brexit. Στις τελευταίες ε, διαπραγματεύσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, είδαμε μια μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μας. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπαρνιέ, τον κύριο Τούς και τον κύριο Γιούνκερ. Ελπίζω ότι θα σκεφτούμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο οι Βρετανοί επέλεξαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. και ελπίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 θα έχουμε εναλλακτικές έναντι των τελωνιακών ελέγχων. Οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισαν μια συμφωνία και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Θέλουν μάλιστα ε, ταχύτατα την δική μας συγκατάθεση και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ε, η 31η Οκτωβρίου είχε καθοριστεί άλλωστε ως ημέρα αποχώρησης όχι από το Βρετανικό λαό αλλά από το ίδιο το Συμβούλιο τον Απρίλιο. Κανείς δεν θέλει παράταση. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι θέλουν να δουν πώς θα, πώς αντιδράσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Όμως το δικό μας έργο είναι τελείως διαφορετικό. Ε, κανείς, ούτε ο κύριος Φερχόφστατ, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αποχώρησης ε, θα εξεταστεί σήμερα από το ε, Κοινοβούλιο, ε, από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Όταν περάσει από εκεί νομίζω ότι αυτό θα είναι το κατάλληλο μήνυμα προς πολλούς από εδώ. Προφανώς κάποια μπλεξίματα μπορούν να γίνουν, να παρουσιαστούν στο μέλλον, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί εμάς. δεν θα πρέπει μέσω αυτού να εκφραστούν άλλες πολιτικές βουλήσεις θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σημαντικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να κάνει ένα ακόμα λάθος ε, χρονική σειρά. Θα πρέπει να τελειώνουμε με τον Brexit. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίρντεναν τώρα έχει το λόγο. Πρόεδρος Σίρντεναν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας ε, αφήνουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά και δεν ε, συνέβαλα στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Αντιθέτως, ε, ε, επιδίνωσαν το προηγούμενο status quo με τη συζήτηση για την ένταξη της Βορείου Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πυροδοτήθηκε μια κυβερνητική κρίση στην Βόρεια Μακεδονία. Ε, όσον αφορά τους ε, κλιματικούς ε, στόχους του 2020 οι ίδιες οι χώρες μέλη δεν ξέρουν τι θα γίνει. Ωστόσο χαίρομαι που το Συμβούλιο υιοθέτησε την πολιτική αξιολόγηση της δικής μου πολιτικής ομάδας ότι η στρατηγική επέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και ο πόλεμος με τους Κούρδους είναι, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, αν το Συμβούλιο και η Κομισιόν αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση, γιατί παραμένουν αδρανείς και δεν επιβάλλουν ε, κυρώσεις. Εμείς είμαστε υπέρ με ενός άμεσου τερματισμού των εξαγών όπλων στην ε, Τουρκία και επίσης ε, μια, είμαστε υπέρ μιας αναγνώρισης της αυτοδιαχείρισης των Κούρδων. Με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουμε θετικά. Τώρα, σχετικά αφορά το Brexit, η δική μου πολιτική ομάδα τις περασμένες εβδομάδες ε, εργάστηκε επικοδημητικά προκειμένου να εξεύρει μια λύση εδώ. Προτεραιότητά μα ήταν πάντα η εξασφάλιση τη ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων εκατομμυρίων πολιτών. Και τώρα υπάρχει ένα νέο deal το οποίο προφανώ αντιμετωπίζει κάποιε δυσκολίε, ε, ε, το οποίο είναι δύσκολο να περάσει από την Βουλή. Εμείς ε, αναμένουμε ένα εγκεκριμένο κείμενο από το Λονδίνο και αυτή στιγμή ε, εκπονηθεί. Θα το αξιολογήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα χρόνο να το κάνουμε. Και αυτή στιγμή ε, υπάρξει αυτό το κείμενο. Θα ήθελα να πω το εξής. Εάν υπερψηφίσετε την παράταση, τότε θα δώσετε τη δυνατότητα στο βρετανικό λαό να λάβει ε, ο ίδιος μία απόφαση. Και ε, κύριε Τούσκ, παρά τις ε, πολιτικές διαφωνίες που είχαμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιονγκιόζη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να περιοριστώ στο ζήτημα του Brexit κάτι το οποίο έχουμε προσπαθήσει να διευθετήσουμε τα τελευταία τρία χρόνια. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει σεβαστό, μόνο ότι το περιθώριο είναι μικρό το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να μπορέσει να αποχωρήσει εφόσον αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κύριο Γιούγκερ όταν είπε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί παράταση. Ανεξάρτητα του αν υπάρχει ή όχι συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποχωρήσει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι προ το συμφέρον τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποχωρήσει δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση που έχουν λάβει οι Βρετανοί πριν από τρία χρόνια δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν. Σαφώ υπήρχε ένα βρετανικό ευρωσκεπτικισμό ήδη από τον Ερίκο τον 8ο και νομίζω ότι αυτό βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά τη ε, γεωπολιτική ε, προσέγγιση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφεί απέναντι στι προτεραιότητέ μα. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πολιτικέ κοινωνικέ ανισότητε, μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει για όλα αυτά να βρούμε μία λύση. Αν η Ευρώπη λοιπόν θέλει να έχει μια επιτυχημένη πολιτική σε όλα αυτά τα σημεία. Αυτά θα πρέπει να καταφέρει να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια και θα πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει όλη αυτή την κόποση που υπάρχει σε σχέση με τη διαδικασία τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να καταφέρουμε επίση να αντιμετωπίσουμε σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο διάφορους που προσπαθούν να παρεμποδίσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί πλέον μια απόφαση και να τελειώνουμε με την ιστορία του Brexit. ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Χούπνερ για δύο λεπτά. Πρόεδρε Τούσκ, Πρόεδρε Γιούνκερ, αγαπητέ Ζων Κλοντ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσήλωσή σας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σχόλια σας για τη διεύρυνση σήμερα. Θα μιλήσω όμως για το Brexit. Ε, τις επόμενες μέρες εμείς εδώ θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη συμφωνία αποχώρησης και να δώσουμε ενδεχομένω συγκατάθεση. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη απρόβλεπτες εξελίξεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πάντως, ε, η δική μας συγκατάθεση θα πρέπει να δοθεί μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Βρετανία. Πράγματι είναι λίγο σαν τεζαβί, διότι και πάλι δεν ξέρουμε τι πλειοψηφίες θα προκύψουν στις διάφορες ψηφοφορίες στη Βουλή των Κοινοτήτων και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε σήμερα τι θα προκύψει από την ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα. Μια ακόμα φορά η διαδικασία χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, όπως και προηγουμένως σε αυτό το μακρύ ταξίδι. Η δεύτερη παράταση τελειώνει αυτή τη στιγμή η μεταβατική περίοδος ε, που προβλέπει η συμφωνία θα μπορούσε να χρησιμεύσει χωρίς άλλη παράταση προκειμένου να προσαρμόσουμε στο καλύτερο τις μελλοντικές μας σχέσει. Να τελειώσω υπογραμμίζοντας ότι ε, η αρνητική κάλυψη των ε, δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, η χρήση δευτερογενούς νομοθεσίας και αυτά που ακούμε από την επαφή μας με τους πολίτες δείχνουν ότι τα δικαιώματά τους ενδεχομένω φοβούνται ότι δεν θα γίνουν σεβαστά στο μέλλον. Ε, όμως τα δικαιώματά τους καθορίζονται και προστατεύονται από τη Συμφωνία Αποχώρησης όταν αυτή επικυρωθεί. Ευχαριστώ. Ο κ. Περέιρα για δύο λεπτά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε μια νέα Συμφωνία Αποχώρησης με το με τη Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτό είναι καλό νέο. Πέραν πάση λογική αμφιβολία, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ως στόχο να δυσκολέψει τη ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαπραγματευθήκαμε μάλιστα συμφωνίε με τρει διαφορετικού πρωθυπουργού. Τον κύριο Κάμερον, την κυρία Μέη και τώρα τον κύριο Τζόνσον. Μια συμφωνία θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε ένα έφτακτο Brexit και να αποφύγουμε τα καταστροφικά σενάρια. Επίσης όμως γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση για αυτή την προτινόμενη συμφωνία. Η θέση του Κοινοβουλίου και της ομάδας μας είναι σαφέστατη. Δεν θα δώσουμε τη συγκατάθεσή μας μέχρι ότου το Βρετανικό Κοινοβούλιο να έχει εγκρίνει τη συμφωνία. Και ας είμαι σαφής. Οποιοδήποτε ψηφοφορία περί συγκατάθεσης έχει σχέση όχι μόνο με την τελική πλειοψηφία στην Ολομέλεια, αλλά και στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Και όταν λέμε έγκριση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, εννοούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βουλή των Λόρδων και η Βουλή των Κοινοτήτων θα πρέπει να έχουν εγκρίνει πρώτα τη συμφωνία. Και όταν λέμε <laughs> ότι η συμφωνία θα πρέπει να έχει εγκριθεί, εννοούμε την τελική επικύρωση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, αφότου θα έχουν συζητηθεί όλες οι προτάσεις τροπολογίας, μεταξύ αυτών και αυτή που ζητά ο λαό να αποφασίσει τελικά με δεύτερο δημοψήφισμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πανέτοιμο, μόλις το Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ψηφίσει και να δώσει την κατάθεσή του. Αν χρειαστεί παράταση, η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Θα στηρίξουμε αυτό το αίτημα. Και στηρίζουμε και τη σημαντική πολιτική δήλωση του κ. Τούσκ σήμερα. Η απόφασή μας δεν θα είναι ποτέ υπέρ μιας αποχώρησης της Βρετανίας χωρίς συμφωνία. Αυτή τη δήλωση τη στηρίζει και η ομάδα μου και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Τώρα για δυόμιση λεπτά ο κύριος Φερχοφστάτ. Καταρχήν, θα ήθελα να πω στον κύριο Βαν Όρντον ότι με τιμά το γεγονός ότι με συγκρίνεται με τον κύριο Πέρκο. Είναι καλύτερο <laughs> από άλλες... Ε, από όταν με συγκρίνουν τον κύριο Ρίσμοκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διάσκεψη των Προέδρων ότι επικύρωσαν ότι η διαδικασία συγκατάθεσης στο σώμα εδώ θα ξεκινήσει μόνο μετά την πλήρη επικύρωση εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας και είναι σημαντικό αυτό να αναφέρεται στα ψηφίσματά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να αξιοποιήσετε το χρόνο από τώρα μέχρι την ε, ψηφοφορία προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία κρεμούν. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαβιούν στη Μεγάλη Βρετανία και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Οι, ε, οι, οι τροτές, οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμών ε, που χρειάζονται συνδρομή και ένα από τα μέλη της Μεγάλης Βρετανίας είπε ότι μπορεί να γίνει εξαγωγή αυτών των ανθρώπων και θα πρέπει να ενταχθούμε ρητά σε αυτό. Ε, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι πλήρως εγκατεστημένοι και αυτοί που βρίσκονται σε ένα προηγούμενο στάδιο. Ε, κατ' εμέ ε, θα πρέπει πραγματικά να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτών των ομάδων. Πριν λοιπόν το σώμα αυτό δώσει τη συγκατάθεσή του, θα ήθελα να επιληθούν αυτά τα προβλήματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, δεν θέλουμε οι πολίτες αυτοί να γίνουν θύματα στην Μεγάλη Βρετανία ενός καινούριου σκανδάλου. Τέλος, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία να πω κάποια θετικά πράγματα για τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ παρόλο που δεν παρευρίσκεται πλέον εδώ. Και επίσης και στον κύριο Τάσκ να, ε, να τον ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και θα ήθελα να του ευχηθώ καλή επιτυχία ε, στις προκλήσεις που τον αναμένουν τώρα σε μια σημαντική χώρα στην ε, Ανατολική Ευρώπη. Καλή τύχη, Ντόναλτ. Για 1,5 λεπτό, κύριο Σμίθε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το Brexit. Δεν θα σας κάνει εντύπωση αυτό. Πρόεδρε Τούσκα, εξ ονόματος της περιφέρειάς μου στη Σκωτία. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω γιατί κρατείτε ανοιχτές τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μας, Είστε ένα πραγματικό φίλο προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Σα ευχαριστώ ειλικρινά γι' αυτό. Την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μιλήσουμε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα πει ότι υπήρχαν ορισμένοι στα πλαίσια τη της Βρετανική κυβέρνηση που α, κακή την πίστη προσπαθούσαν ουσιαστικά να απορρίψουν οποιαδήποτε συμφωνία εσείς διαπραγματευόσασταν καλή την πίστη. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ γρήγορα είδαμε ότι γινόντουσαν διάφορες γρήγορες κινήσεις προκειμένου να καταρριφθούν κάποιες αποφάσεις προστασίας των επιχειρηματιών ή των αυτοαπασχολούμενων δευτέρων επαγγελματιών που κατοικούν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρομαι σε Ευρωπαίου πολίτε. Του δόθηκαν διάφορε εγγυήσει ότι τίποτα δεν επρόκειτο να αλλάξει προ το καθεστώ του. Οι άνθρωποι όμω αυτοί περιμένουν ακόμα την διασφάλιση αυτή μέχρι να εγκριθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καθεστώ χάου από μία λεπτή κλωστή κρέμετη κυβέρνηση του Μπόρι Τζόνσον. Πραγματικά δεν μπορούμε να του εμπιστευτούμε ακόμα και αν δείξουν καλόπιστη προσήλωση συμφωνία αυτή. Μάλιστα έχουμε μία επιστολή από τους πρωθυπουργούς της Σκοτίας και της Ουαλίας θεωρώ ότι και εμεί θα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα. Προβλέπεται επίσημη συγκατάθεση και από τα δικά μα τοπικά κοινοβούλια. Εμεί δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δώσουμε μια τέτοια έγκριση και σίγουρα αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται το Βρετανικό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει διαδικασία ανάλυση και επικύρωση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε εμεί τα δικά μα τοπικά κοινοβούλια να είναι συνένοχα στην πολύ άσχημη αυτή κατάσταση που έχει προκύψει. Σίγουρα ο χρόνος γιατρεύει πάρα πολλά πράγματα και η παράταση αυτή η οποία έχει ζητηθεί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί τώρα για ένα χρόνο, για μεγαλύτερο ακόμα χρονικό διάστημα ο κύριος Τζόνσον ενδεχομένω να έχει σπαταλήσει άδικα το χρόνο αυτό. Εμείς θα αξιοποιήσουμε τον νέο χρόνο που ελπίζω να μας δώσετε προκειμένου να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλην χρησιμοποίησε περισσότερο χρόνο από ό,τι σου αναλογούσε. Ήμουνα υπομονετική γιατί έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, αλλά σα παρακαλώ πολύ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσή σα. Για ένα λεπτό, ο κύριο Μόιτεν έχει το λόγο. Κύριε ε, Πρόεδρε, κύριε Τούσκ, ε, κύριε Γιούγκερ, ε, ζούμε μια συνεχή φάρσα. Οι Βρετανοί με πλειοψηφία αποφάσισαν υπέρ μιας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκάθαρα. Αλλά μέχρι τώρα κανένα αποτέλεσμα. Ε, ποιος θέλουμε να εξηγήσει στους πολίτες πώς ε, υπονομεύεται η επικύρωση της Συμφωνίας ε, Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήστε να κάνετε τη συμφωνία αυτή καθόλου ελκυστική, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εμείς περιμένουμε μαζί με τον κύριο Πέρκο να γίνεται μία επαόριστον αναβολή αυτής της εξόδου. Είναι ένα θλιβερό θέαμα. Εγώ το παρακολουθώ κλαίγοντας και γελώντας ταυτόχρονα. Ε, κλαίγοντας γιατί είμαστε ιστορικοί μάρτυρες του πώς διαστρεβλώνουν δημοκρατικές διαδικασίες. Γελώντας γιατί υπάρχουν ε, μέλη του κόμματος του Brexit των οποίων τα νεύρα είναι τεντωμένα και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερος. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Άνσεπ. όχι, δεν ήταν μπλε κάρτα, σας ζητώ συγγνώμη. Άρα δεν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα μέσω μπλε κάρτας. Όχι. Περνάμε τότε στον κύριο Έπινγκ για ένα λεπτό ευθύ αμέσω. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κατάφερε να εγκρίνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Και ευτυχώς, ευτυχώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γαλλία. Δεν προβλέπεται ακόμα προσχώρηση των ε, χωρών αυτών. Φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα Βαλκάνια. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πολύ ευτυχή εξέλιξη. Στην Αλβανία τεράστιο επίπεδο διαφθοράς. Ίδιο επίπεδο με τον Παναμά και την Κολομβία. Δείτε λίγο τη Ρουμανία που ήταν το 2007. Όλοι νομίζαν τότε ότι η Ρουμανία ήταν έτοιμη για ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφθορά ήταν σημαντικότατο πρόβλημα τότε. Υπήρχαν χρηματικέ ε, ροέ προ την Ρουμανία παράνομε και παρόλα αυτά η χώρα αυτή εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτοτε έχουμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να δημιουργεί το τέρας το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, δηλαδή την ηγεμονία Ερντογάν. Η Γαλλία νομίζω ότι κράτησε πάρα πολύ σωστή στάση απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία. Δεν συμφωνώ πάντα με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά έχω να του πω αυτή τη φορά merci beaucoup. Okay. Κύριε ε, το Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθεί να είναι ε, πραγματικότητα. Ε, και αν δώσουν βέτο στους ενωτικούς, ποτέ δεν θα ξανασυγκαλυθεί η συνέλευση του Στόρμοντ. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία και επιτρέπει ένα κοινό καθεστώς ε, για τα αγαθά στην Ιρλανδία. Ε, όμως ε, τα εργατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το η περιβαλλοντική προστασία θα είναι χαμηλότερη για την Ιρλανδία. θα είναι μέσα στην Ευρώ, στο ευρωπαϊκό σπίτι, αλλά θα είναι και έξω από το ευρωπαϊκό σπίτι η Βόρειο Ιρλανδία. Αυτό δεν θα είναι πολύ καλό. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να προγραμματίσουμε για την Ιρλανδική ενότητα, όχι να μείνουμε ε, σκλάβοι μιας ε, συμφωνίας. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρης το λόγο. Το κουμπάκι είναι μπροστά σας για να ανοίξει το μικρόφωνο. Οι α, βουλευτές στο δικό μου το κοινοβούλιο σταματάνε αυτή τη στιγμή μια συμφωνία την οποία την έχουν ζητήσει οι Βρετανοί πολίτες δεν νομίζω ότι πρέπει ή μπορούμε να κυρώσουμε το Brexit. Δεν υπάρχει μια εντολή για τους βουλευτές για να κάνουν κάτι τέτοιο. Έχουμε χάσει τον έλεγχο. Οι άνθρωποι στη δική μου την περιφέρεια έχουν χάσει τον έλεγχο που θα πρέπει να έχουν. Δεν εγκαταλείπουμε όμως. Οι περισσότεροι Βρετανοί θέλουν να τροποποιήσουν το αποτέλεσμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εκατομμύρια ψηφοφόροι οι οποίοι εκφράστηκαν το 2016 σαφώς και δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια αυτή. Δείχνουν την καλύτερη εικόνα των Βρετανών μέσω της αιμονής τους απέναντι σε όλες αυτές τις αντικσότητες. Ενδεχομένως να προσπαθήσετε να μας αποδυναμώσετε μέσω όλων αυτών των διαφορετικών διακυμάνσεων των διαπραγματεύσεων, αλλά εγώ πάντως πιστεύω ότι η δική μας η θέληση δεν μπορεί με τίποτα πραγματικά να νικηθεί. Η φωνή των πολιτών θα ακουστεί. Κυρία Χάρης, κυρία Χάρης, μ' ακούτε? Η πρόεδρος προσπαθεί να μιλήσει μαζί σας. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από την κυρία Γραπίνη, μα λατρεύω τις συζητήσεις, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γραπίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε, στην παρέμβασή σας μας δώσατε και μία πληροφορία. Είπατε ότι η πλειοψηφία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θέλουν να αλλάξουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Από πού προκύπτει αυτή η πληροφορία, γιατί εμείς τέτοια πληροφόρηση δεν λάβαμε. Το αντίθετο μας λένε ότι οι περισσότεροι Βρετανοί πολίτες θέλουν τώρα να αλλάξουν ε, την απόφαση του δημοψηφίσματος. Από πού προκύπτει λοιπόν η πληροφόρησή σας αυτή. Ένα 54% φαίνεται ότι είναι υπέρα της αποχώρησης, και ας μην ξεχνάμε τα 17 εκατομμύρια που ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης το 2016 εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία. Το 54% προκύπτει από μια πρόσφατη δημοσκόπηση προηγούμενης εβδομάδας. Η κυρία Φόρντεν θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. να σας υπενθυμίσω ότι το σλόγγαν που χρησιμοποιήσετε το 2016 ήταν «Take back control», να κτίσουμε τον έλεγχο. Με αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το κοινοβουλίο μας. Αυτό δεν θέλετε κι εσείς. Στη δική μου τη χώρα οι άνθρωποι είναι κυριαρχοί. Στη δική μου τη χώρα οι ε, πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την νομοθεσία μας. Το κόμμα του Brexit είναι πάρα πολύ νέο. Δεν υπήρχε το σλόγγαν αυτό τότε. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Γκιόρη έχει το λόγο. Κυρία Γκιόρη, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ορισμένοι αρχηγοί κρατών Δυστυχώ δεν μπορούν να σκεφτούν με μια μακροπρόθεσμα προεπτική. Αυτό μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε πρόσφατα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσει με την ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Εμείς χώρες του Βίζενγκρατ, είπαμε ότι η απόφαση αυτή υπονομεύει την αξιοπιστία μα και έχει δυσμενεί επιπτώσει στη δική μα ε, σταθερότητα θα πρέπει να υπάρξει μια γεωπολιτική ε, ε, σταθερότητα ε, που δεν είναι πλέον εφικτή γιατί οι χώρες αυτές δεν μπορούν να έρθουν πιο κοντά μας. Μεταθέτουμε αυτό το στόχο, χάνουμε την αξιοπιστία μας και δεν θα πρέπει να τρέφουμε πλέον ψευδεστήσεις θα έχουμε κάποιους ανταγωνιστές οι οποίοι θα μπορέσουν να σκεφτούν πιο μακροπρόθεσμα και θα έρθουν να καλύψουν το κενό που δημιουργήσαμε εμείς. Τέλος, είναι πολύ αξιοσημείωτο το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα που έχουμε διαψεύσει δύο ευρωπαϊκές ε, χώρες, κανείς ε, δεν είπε ότι αυτοί οι οποίοι μπλοκάρισαν την ένταξη αυτών των χωρών δεν είναι γνήσιοι ευρωπαϊστές, ενώ το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλες περιπτώσεις. Κυρία Φρίτσον, για ένα λεπτό. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την τροποποιημένη συμφωνία ε, αποχώρησης και μια πολιτική δήλωση. Από την ε, ευρωπαϊκή πλευρά έχουν γίνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μια συμφωνία θα είναι εφικτή για να αποφύγουμε ε, την έξοδο της Βρετανίας χωρίς συμφωνία. Και ο Μισελ Μπαρνιέ πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να τον συγχαρούμε κατάφερε να διατηρήσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονό ότι η Βρετανία βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας ανησυχεί, αλλά σεβόμαστε την ε, επιθυμία του Βρετανικού λαού. Υπάρχουν Βρετανοί που ζητούν ένα δεύτερο δημοψήφισμα και εν πάση περιπτώσει ο Μπόρις Τζόνσον έχει πολύ μεγάλη και βαριά ε, την ευθύνη στους ώμους του. Ελπίζω ότι θα βρούνε έναν τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you. One minute. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Πόριτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ τους Ευρωπαίους φίλους μας ε, που εξακολουθούν να ε, υπομένουν, να δείχνουν υπομονή. Αυτή η συμφωνία είναι μια ορλαϊκή βόμβα. Αν περάσει και από την Βρετανία και από το Κοινοβούλιο, σε ένα χρόνο περίπου θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα είναι πολύ κοντά στη μη συμφωνία. Γιατί τα εργασιακά δικαιώματα, η φορολογία, η περιβαλλοντική προστασία, όλα αυτά θα πληγούν. Γιατί όλα αυτά έχουν βγει από την συμφωνία και έχουν μπει στην πολιτική δήλωση. Ε, και αν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ Βετανίας και Ευρώπης ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πολύ δύσκολο αυτέ οι, οι, για τη μελλοντική εμπορική σχέση να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο. Οπότε, δεν θα έπρεπε να υποθηκεύσουμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των νέων στο μέλλον, των εργατών κλπ. Ο πρόεδρος Τούσκ αναγνώρισε την ανάγκη ε, να, την, ε, την ενδεχόμενη ανάγκη να δοθεί μια καινούρια ε, παράταση και θα πρέπει να τη δεχτούμε. Ευχαριστώ. One minute now for Madam Phillips. Ένα, ένα λεπτό για την κυρία Φίλιπς. Σα Σας ευχαριστώ. Το Σάββατο συμμετείχα και εγώ στη διαδήλωση των εκατομμυρίων ανθρώπων στο Λονδίνο ζητώντας ένα νέο δημοψήφισμα γιατί πιστεύω ότι το να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη διεφθαρμένη αυτή συμφωνίας του Μένου Βασιλείου ουσιαστικά αποδυναμώνει την κατάστασή μα τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντο. και πραγματικά θίγει πάρα πολλέ κοινότητε, οι οποίε είναι εγκαταλειμμένε εδώ και ολόκληρε δεκαετίες από την Βρετανική κυβέρνηση. Η συμφωνία αυτή θα επηράσει το σύνολο τη επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είναι οι πιο ομάδε, όπω οι γυναίκε οι οποίοι επηρεαστούν περισσότερο οι έγχρωμοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε ένα νέο δημοψήφισμα, προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να επιλέξουμε ανάμεσα στη συγκεκριμένη αυτή συμφωνία και τη δυνατότητα παραμονής τον Ιούνιο του 2016 δεν πέθανε η δημοκρατία και υπάρχει ακόμα μια πλειοψηφία στην ε, χώρα μας που θέλει κάτι το διαφορετικό, κάτι διαφορετικό. Επομένως αυτό το οποίο λέω εδώ πέρα στο Στρασβούργο, απευθυνόμενοι προς τη χώρα μου, δεν πρόκειται να καταλήψω τους εργαζομένους, το περιβάλλον και όλους εκείνους που θα φυγούν από την επικίνδυνη αυτή συμφωνία. Δεν πρόκειται να καταλήψω την προσπάθεια και να παραμείνει τον Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε δύο μπλε αν όχι τέσσερις. Δέχεστε. You don't have to, but it's your choice. Δεν είστε υποχρεωμένοι. Μπορείτε να το επιλέξετε. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Mr. Habib. Yeah. Habib, έχει το λόγο. Habib. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φίλιπς ε, αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη μείωση των προτύπων αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύει, δεν έχει την παραμικρή αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ακόμα και κατανόηση των βασικών βρετανικών αξιών που διέπουν τη χώρα μας, αλλά και όλο τον πλανήτη για το καλό της ανθρωπότητας, αλλά και την ελευθερία της χώρας μας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί. Ας ακούσουμε και την απάντηση. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι συνάδελφοι εκεί απέναντι φοβούνται τόσο πολύ τη δημοκρατία και για ποιο λόγο δεν δίνει τη δυνατότητα πάλι στους πολίτες να αποφανθούν για κάτι το οποίο θα πειράσει το δικό τους το μέλλον αλλά και το μέλλον όλης της Υπήρου. Σας ευχαριστώ. I might actually run clapometer on the next question that comes from Mr. Foreman. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Φόρμαν δύο μπλε μόνο κάρτες. Δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερις ερωτήσεις. The lady. Ε, προς την συναδελφό σας θα θέσετε το ερώτημα. Κύριε Φόρμαν, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε την ερώτησή σας. Μα τη δεχθήκατε ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά δεν ρώτησα πρώτα την συνάδελφο αν θα ήθελε να απαντήσει και είπε ότι δεν θέλει να απαντήσει σε ενδεχόμενη ερώτησή σας. Άρα Προχωράμε στον επόμενο εγγεγραμμένο μιλητή που νομίζω ότι είναι ο κύριος Καμπομενόζη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποιος πριν από λίγο είπε ότι έχουμε έναν ντεζαβού σε σχέση με τη συζήτηση αυτό, μα αυτό αληθεύει απόλυτα. Πριν από δύο χρόνια νομίζαμε ότι η συμφωνία για το Brexit θα εγκρινότανε αλλά νομίζω ότι το ότι δεν έχει εγκριθεί δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο με τα σφάλματα τα οποία έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία, μια τροποποιημένη συμφωνία. Θα δούμε αν αυτή θα γίνει τελικά αποδεκτή, θα δούμε που θα οδηγήσει. Το πρόβλημα όμω είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο πλανήτη είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Σαφώς δεν είναι προβεβλημένη στο διεθνές προσκήνιο. Και πολλές φορές χρησιμοποιεί τις διεθνείς κρίσεις προς το δικό της συμφέρον. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησε το δημοψήφισμα στη Σκοτία για να αποσταθεροποιήσει τον Αμένο Βασίλειο, αγνοεί εντελώς συνειδητά όμως τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καταλωνία. Νομίζω ότι σε ζητήματα όπως το Brexit θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ο κύριος Λούνγκρεν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση πραγματικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η χώρα γίνεται όλο και λιγότερο δημοκρατική και υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες και η συμβίωση επαπειλείται θα πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η, η Τουρκία έχει η ίδια δυσφημίσει τον εαυτό της. Όταν μιλούμε για τον προπολογισμό, εδώ θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως μια αναγκαία περικοπή. Αλλά θα πρέπει να δούμε το εξής. Στη δική μου χώρα, την Σουηδία, 50 δισεκατομμύρια κορώνες ε, καταβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε είμαστε ένας από τους πιο σημαντικούς καθαρούς ε, πληρωτές. Και αντί τούτου τώρα διεξάγεται μια συζήτηση ε, σε σχέση με το τι μπορούμε να πάρουμε πίσω. Ε, τι γίνεται με τις εμπορικές ροές. Αυτές είναι σημαντικές. Για ένα λεπτό, κύριος Κάρθη. Τα σύνορα είναι ήδη πολύ σκληρά και δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας και πολύ πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα. Η Συμφωνία της Μεγάλης ε, Παρασκευής ήταν τα εργαλεία για να αποζημιωθούμε για τις βλάβες των περασμένων δεκαετιών. Γι' αυτό το Brexit ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη ε, εξέλιξη, γιατί υπονομεύει την οικονομία της ε, Ιρλανδίας και θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα σε σχέση με τα σύνορα. Εμείς τα υποστηρίξαμε γιατί είναι καλύτερο από την εναλλακτική δυνατότητα, αλλά συμφωνία δεν μπορεί να αποδυναμωθεί. Δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρξουν ευκαιρίες ε, για να γίνουν οικονομικές ε, συναλλαγές. η δυνατότητα του βέτο είναι παραπλανητική. Η μόνη δυνατή προστασία της χώρας μας είναι μέσω μιας ενωμένης Ιρλανδίας και ελπίζω ότι το σώμα αυτό θα είναι διατεθειμένο να, στην, να διεξάγει την μεγάλη συζήτηση. Για ένα λεπτό, κύριο Αλαβάνος έχει το λόγο. Είναι επικίνδυνε για τους λαούς οι αποφάσει του Συμβουλίου που αποτυπώνουν μεγάλες αντιθέσεις εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος των σκληρών ανταγωνισμών της με τις Ηνωμένες και τη Ρωσία για το ποιοι όμιλοι θα ωφεληθούν στη συρία αλλά και στα βαλκάνια. η αναγνώριση της τουρκίας σαν ουσιαστικό συνεταίρο σύμμαχη χώρα του νάτο με δίθεν κυρώσει σε μελλοντικού εξοπλισμού, ενώ αυτή εισβάλλει στη συρία τα λένε όλα. Ανάλογε κυρώσει χάδια προβλέπονται για τις τουρκικές παραβιάσεις στο αιγαίο τι γεωτρήσει στην κυπριακή αόζ. το μπλοκάρισμα των ενταξιακών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων με τη βόρεια μακεδονία και την αλβανία φανερώνει μεταξύ άλλων την επιδίωξη της αστικής τάξης της γαλλίας να κερδίσει χρόνο για να αναβαθμίσει το δικό της ρόλο στα βαλκάνια πάντα στο πλαίσιο όμως της επιζήμιας για τους λαούς της περιοχής συμφωνίας των πρεσπών. ο εφησυχασμός και εξοραϊσμός των υπεριαλιστικών συμμαχιών και συμφωνιών από την κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας αλλά και το σύριζα είναι αβάσιμη, είναι επικίνδυνη για το λαό μας ο οποίος πρέπει να επαγρυπνά με την πάλη του ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια. Κύριος πώς έχει το λόγο. Αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε περάσει τουλάχιστον 15 κρίσεις. Μεταναστευτικό, κρίση του ευρώ, την ελληνική κρίση, το Brexit, την ε, επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, το δίζελ, ε, κλιματική κρίση, λαϊκισμός, ε, κρίση του κράτους δικαίου σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομοποίησης ε, των ε, οργάνων ε, και των διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Spitzenkandidaten, τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Brexit που είναι η μεγαλύτερη κρίση, η απόπειρα λαϊκιστικού πραξικοπήματος στην Ισπανία και λοιπά. Πέντε χρόνια Ζωάν Κλώτ πολύ δύσκολα όμως οι 27 είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και πιο ισχυροί από ποτέ. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η πιο καλή πολιτική εφεύρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ε, βλέπω τον Μιγγέλ, τον Μισελ, τον Ιωάννες, ε, ε, όσο δύσκολοι και αν είναι οι καιροί που, θα μας, που μας περιμένουν, έχουμε ένα παράδειγμα από το παρελθόν. Μπορούμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με ενότητα και με αγάπη για το ευρωπαϊκό κατάφερε ένας ε, νότιος όπως εγώ να αισθάνεται Σε Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόρμπετ τώρα έχει το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε θόρυβο. Γιατί πραγματικά δεν δείχνετε κανένα σεβασμό προς τους ομιλητές. Ο κύριος Κόρμπετ λοιπόν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Και ακούστε σας παρακαλώ πολύ τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί αυτή τη στιγμή να περάσει τη συμφωνία αυτή στην Βουλή των Κοινοτήτων μέσα σε τρεις ημέρες, όπου θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή αλλά και στις επιμέρους επιτροπές. Έχουμε μια συμφωνία 110 σελίδων όσον αφορά τους φαρμαστικούς νόμους. Έχουμε την αρχική συμφωνία που είναι 600 σελίδων. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι ε, θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να εγκρίνουμε τη συμφωνία με την υφιστάμενη μορφή της. Σίγουρα θα υποβληθούν τροπολογίες. Ορισμένες τροπολογίες θα έχουν ως στόχο ένα πιο ήπιο Brexit γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολύ σκληρό Brexit που βγάζει το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός εσωτερικής αγοράς, εκτός Τελωνιακής Ένωσης, θα βλάψει την Βρετανική αλλά και την Ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι κακή συμφωνία τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υποβληθούν όμω και κάποιε τροπολογίε, σύμφωνα με τι οποίε θα πρέπει να αποφανθεί πάλι ο Βρετανικό λαό για οποιαδήποτε αποχώρηση και αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό γιατί το ενδεχόμενο αποχώρηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα με ένα τέτοιο τρόπο που διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που είχαμε πει στου πολίτε όταν ψήφισαν για πρώτη φορά το 2016. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτε που θέλουν εκ νέου να αποφανθούν. Το λένε αυτό ξεκάθαρα και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στι διαδηλώσει που έλαβαν χώρα στο Λονδίνο. Και αυτό δείχνουν και περισσότερε δημοσκοπήσεις. Ότι ο Βρετανικό λαό θέλει και του αξίζει να αποφανθεί εκ νέου για την καταστροφική αυτή απόφαση για τη χώρα πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κόρμπετ, δύο μπλε κάρτες έχουν υποβληθεί. Μπορώ να δεχθώ μία μόνο, γιατί ήδη έχουν εγγραφεί 20 ομιλητές στη διαδικασία Catch the Eye. Δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Ντόγκνε. Ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας. Κύριε Ντόμπνε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τον κύριο Κόρμπετ το ακόλουθο. Τι θα έλεγε στα 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους των εργατικών και στο 60% των εργατικών που ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείτε να τους πείτε ότι δεν προδίδετε εσείς τη στάση τους τη στιγμή που εσείς αυτή τη στιγμή, όντας σοσιαλιστής, ζητάτε να διεξαχθεί δεύτερο δημοψήφισμα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Απάντηση οι περισσότεροι ψηφοφόροι των εργατικών ήταν υπέρ της παραμονής κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος και είχε αυξηθεί αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους γιατί ακόμα και αυτοί που ψήφισαν αρχικά υπέρ της αποχώρησης είδαν ότι όλη η διαδικασία τους Brexit είναι μια ακροδεξιά ουσιαστικά διαδικασία που υποστηρίζεται από τις πιο σκληρές πτέρυγες των Tories που πραγματικά θα στραφεί κατά της οικονομίας μας των θέσεων απασχόλησης και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ωφελεί το Μένο Βασίλειο. Γι' αυτό το λόγο το εργατικό κίνημα, το εργατικό κόμμα με συγχωρείτε πλέον πιστεύει ότι οποιαδήποτε απόφαση κι αν ληφθεί θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγηση από το Βρετανικό λαό εκ νέου μέσω δεύτερου δημοψηφίσματος. Ο κύριο Κέλιχερ έχει το λόγο. Εξ αρχή θα ήθελα να πω ότι αποδέχομαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί που ήταν υπέρ τη αποχώρησης αυτής σε καμία περίπτωση δεν θα θέλανε ένα σκληρό Brexit, Χωρί συμφωνία δηλαδή, το οποίο σίγουρα θα στραφεί κατά τη κατάσταση στην Βόρεια Ιρλανδία και τη ίδια τη συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή έχει γίνει κέριο και ακαθόδε ζήτημα στι συζητήσει που γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασίλειου. Είμαστε όμω σαφέστατοι. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η οποία παρεμποδίζει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το ίδιο το Βρετανικό το Κοινοβούλιο που έχει εμπλακεί σε μια πολύπλοκη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει βέβαια να συνάδει με την αρχική συμφωνία, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ίσο της Ιρλανδίας. Υποτίθεται ότι η συμφωνία αυτή θέλει να την προστατεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η απαραίτητη δημοκρατική λογοδοσία στην Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά και βέβαια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μειώσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στη στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Ιρλανδία, θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν εκεί. Θα είναι πραγματικά στο αν διώξουμε του Ευρωπαίου πολίτε από την Βόρεια Ιρλανδία. Η κυρία Ράιντεκε έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αφηγούνται, αφηγούνται μια ιστερία στην ε, Μεγάλη Βρετανία ε, ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κουραστεί από εμά, θέλουν να μα ξεφορτωθούν. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό το κοινοβούλιο είναι και το κοινοβούλιο των Βρετανών υπηκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κουραστεί από τη Μεγάλη Βρετανία ούτε από του Βρετανού πολίτε. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κουραστεί από λογικές διαπραγματεύσει. Εμείς αγαπούμε τις διαπραγματεύσει και την εξέβρεση κοινών λύσεων. Αυτό το οποίο μα έχει κουράσει είναι οι πρωθυπουργοί οι οποίοι δίνουν, εξαγγέλουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τηρήσουν και χρησιμοποιούν υποκριτική γλώσσα σε τέτοιες συγκυρίες. Ε, ε, μας έχουν κουράσει οι πρωθυπουργοί που δεν κατανοούν ότι στην περίπτωση που δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία από τη Βουλή Κοινοτήτων θα πρέπει να γίνει ένα διποψήφισμα ώστε οι Βρετανοί πολίτες να μπορούν να αποφασίσουν ήδη τελικά και οριστικά. Mr. Madison, for minute. κύριος Μάντισον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με πολλά πράγματα με τον κύριο Γιούγκερ, αλλά όπως είπε πριν από πέντε μέρες δεν υπάρχουν επιχειρήματα για μια περαιτέρω παράταση. Για τους συναδέλφους από την αριστερά που αναφέρονται στην δημοκρατία, για τους φόβους για ένα νέο δημοψήφισμα, θα ήθελα να πω ότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν εκατομμύρια πολίτε που δεν ικανοποιούν από το γεγονό ότι βρίσκεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε νέε ευρωεκλογέ, γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ε, εκλογών. Βεβαίως όχι. Το ίδιο θα ισχύει και για ένα νέο δημοψήφισμα, ίσως σε 10-20 χρόνια. Θα υπάρξει ένα νέο δημοψήφισμα ένταξης, επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η συντηρητικη η δεξί τόρις, ε, δεν θα, δεν, θα κερδίσουν τι επόμενε εκλογέ επειδή έχουν ολοκληρώσει το Brexit. Χάναν, το θέμα δεν είναι η ανηλικρίνεια των βουλευτών, αλλά ε, και το, το, η ευφυΐα τους. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν αρνηθεί το Brexit. Όμως επανειλημμένως ε, είπαν ψέματα και απέκρυψαν τα πραγματικά τους κίνητρα. Πιστεύουν ότι καλώντα συνεχώ για εκλογέ αλλά ψηφίζοντα εναντίον δεν θα το προσέξουμε. Ε, ότι θα τροποποιήσουν συμφωνία με στόχο ώστε να μείνει η ίδια στην πραγματικότητα ε, δεν θα το προσέξουμε. Και κάθε φορά κάνουν λάθο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συντηρητικοί ε, βρίσκονται σε διψήφια νούμερα και αυξάνουν τη δύναμή τους. Έτσι λένε οι έρευνες. Οπότε ή θα βγούμε τώρα με το ε, Brexit ε, με αυτή τη συμφωνία ή οι συντηρητικοί θα κερδίσουμε μεγαλύτερη πλειοψηφία σε επόμενες εκλογές. Κύριε Σμιθ, μπλε κάρτα. Ε, καταλαβαίνω τις κριτικές για την ανηλεκρίνεια. Ε, ο, ο ίδιος ε, είχε πει κάποτε ότι κανένα δεν μιλάει για αποχώρηση από την ενή αγορά όμως Άρα λοιπόν πως μιλούσε για τον εαυτό του για την κλήρια. επίσης τα δικαιώματα των, των Βρετανών πολιτών δεν θα είναι πια τα ίδια. μήπως θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη και γι' αυτό, γιατί λέγατε ότι θα είναι. Δεν είναι αλήθεια ότι είπα τέτοια πράγματα εγώ κατά διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ε, αυτά τα λέτε από μια συνέντευξη του 2015 πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Και είχα πει ότι ε, το ελβετικό σύστημα θα ήταν το καλύτερο για μας. Εγώ δεν άλλαξα τη θέση μου. Εσείς στηρίξατε όλη σας την καριέρα το ότι ζητούσατε δημοψήφισμα για ένα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα δεν δέχεστε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το οποίο ψήφισε όλος ο Βρετανικός λαός. Θα περάσω στον επόμενο μιλητή. Δεν δεχόμαστε πάνω από μία μπλε κάρτα. Και ίσω αργότερα δεν θα δέχουμε καμία μπλε κάρτα, διότι έχουμε το Catch the Eye. Ο κ. Φαρατζέ, λεπτό. Μετά από τρία χρόνια αγωνιωδών διαπραγματεύσεων, Μισελ Μπαρνιέ κατάφερε τον Μπόρις Τζόνσον να υπογράψει μια καινούργια συμφωνία που εγγυάται τρία ακόμα χρόνια αγωνίας, διαπραγματεύσεων, αγωνιωδών διαπραγματεύσεων που θα μας καταστήσει απικία, καταστήσουν απικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γιατί το κάνει ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί δεν θέλει άλλη παράταση, γιατί ξέρει ότι οποιαδήποτε παράταση θα βλάψει το συντηρητικό κόμμα στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό το λόγο θέλει να υπογράψει συμφωνία πριν ξυπνήσουμε. Το ίδιο έχει συμβεί και στο παρελθόν. Οι Tories ε, βάζουν το συμφέρον τους πάνω από το συμφέρον της χώρας. Εμείς θέλουμε μια συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων που θέλουν να αποσυρθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατέβουμε μαζί στις εκλογές. Μόνο με ένα ξεκάθαρο Brexit μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ. Ε, ήμουν για 20 χρόνια. Λυπάμαι, λυπάμαι που θα σας αφήσω. Θα μ' άρεσε να παραμείνω Φοβάμαι όμω δυστυχώ ότι θα ξανάρθουμε τον Νοέμβρη εδώ πέρα. Εγώ ήθελα να είναι η τελευταία μου ομιλία, αλλά ίσω να μην τα καταφέρω. Στο συγγνώμη, δεν ακούσαμε το τελευταίο τμήμα τη ομιλία του κύριου Φαράζ γιατί φωνασκούσατε. Α ακούσουμε τώρα τον κύριο Ταγιάννη για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλτ, αγαπητέ Ζαν Κλοντ, συμμερίζομαι την απογοήτευσή σας ε, για την μία απόφαση τελικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η Κίνα, η Ρωσία, η Σοδική Αραβία επενδύουν όλο και περισσότερους πόρους στα Βαλκάνια και εμείς οπισθοδρομούμε αυτή τη στιγμή, δεν συμβάλλουμε στη σταθερότητα της Βαλκανικής ε, περιοχής, πράγμα το οποίο θα ήταν πάρα πολύ θετικό για το σύνολο της Ευρώπης. Στέλνουμε τελικά αρνητικά μηνύματα και πραγματικά θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο καταστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο αδιάφορη και αμέτωχη για όλη αυτή την ε, περιφέρεια των Βαλκανίων. Και πρέπει επίση ξεκάθαρα προς τη Μέση Ανατολή να μιλήσουμε προς την Τουρκία, λέγοντας ότι θα πρέπει σε καμία περίπτωση βέβαια να εισβάλλει στην ε, Συρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να συλλάβει τους Κούρδους τρομοκράτες στη δική της την επικράτεια η Τουρκία και όχι να εισβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο σε τμήμα της Συρίας. Εξακολουθούμε πάντως και κάνουμε λάθη αυτή τη στιγμή γιατί λόγω των εθνικών μας εγωισμών δεν καταφέρνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε στο διεθνές προσκήνιο. Δεν είχαμε το θάρρος να απευθυνθούμε στην Τουρκία ή ακόμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου προκειμένου να καταδικάσουμε τις κρατικές ενισχύσεις ενισχύσεις προς τη βιομηχανία χάλιβα της Τουρκίας που ε, συναγωνίζεται με τρόπο αθέμητο την αντίστοιχη ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε πλέον την εθνικιστική μας ε, στάση και να καταφέρουμε πραγματικά να μιλήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πολιτική. Αν η Ευρώπη δεν επιστρέψει σε μια υγιή πολιτική, τότε τι επόμενε δεκαετίε η στάση θα θεωρείται από τι υπόλοιπε χώρε όλο και πιο αδιάφορη. Η κυρία Μάρκε έχει το λόγο. Θέλω να πω δύο λόγια για τον κύριο Γιούνκερ καταρχήν γιατί κατά τη διάρκεια όλης της θητείας του σεβάστηκε την αρχή ε, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αντικατοπτρίζουν όμως τις διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών ε, δεδομένης πρότασης της Φιλανδικής Προεδρίας. Μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών διαφωνούν με την Προεδρία η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε πρόσφατα. Επίσης δεν λαμβάνει υπόψη τη συστάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές ε, προτεραιότητες της ε, νέας Πρόεδρου της Κομισιόν. Οπότε αυτή η πρόταση υστερεί έναντι αυτών που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα 7 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως θα εξακολουθήσει να ασκεί τις αρμόδιτες του και θα διαπραγματευτεί ένα πιο ισχυρό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε προκειμένου να υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να δεχτούμε ένα οποιοδήποτε προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τούσκα, ε, πετύχατε μία συμφωνία με τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ, τον οποίο θα ήθελα να χαιρετήσω σεβόμενοι τους ευρωπαϊκούς κανόνες, επίσης την ε, κυρίαρχη επιλογή του Βρετανικού λαού και θα ήθελα να καταγγείλω εδώ τη στάση του κυρίου Φάρατζ. 20 χρόνια μάχης κατά της Ευρώπης, 20 χρόνια κατά τα οποία αυτός ε, τράφηκε από την Ευρώπη. Σημαντικό σήμερα, σημαντικό σήμερα είναι το μέλλον οι μελλοντικέ σχέσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρνιέ για τα όσα έκανε υπέρ της ε, συνοχής των 27 ε, χωρών προκειμένου να διατηρηθεί ένα όραμα ε, και να, ε, να εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό μέλλον. Ε, Μία νέα αναβολή δεν θα πρέπει να εγκριθεί παρά μόνο αν υπάρξει από χρόνο λόγος νέο στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειες για να εγγυηθείτε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό η κυρία Σκότ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που ο Τζόνσον κάνει τις δικές του προσπάθειες, εμείς προσπαθούμε να εργαστούμε έντιμα προσπαθώντας να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση. Ε, το Brexit ε, δεν θα πρέπει να είναι ένα πλήγμα ε, κατά της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Χαιρετίζουμε την ιδέα του κυρίου Μπαρνιέ για ισότιμους όρους προ... εμποδίζοντας το... τη Μεγάλη Βρετανία να υπονομεύσει την κοινή αγορά και το φορολογικό μας σύστημα. Αλλά τις μέρες αυτές ο κ. Τζόνσον προέβη προς μια πολιτική δήλωση η οποία δεν θα είναι νομικά δεσμευτική και είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι ε, προετοιμάζει τη Μεγάλη Βρετανία να γίνει μια απειλή όσον αφορά την ακαιρεότητα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ότι δεν θα εγκρίνουμε τη συμφωνία πριν από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να επιμείνουμε εδώ παρά τις πιέσεις που μπορούν να προέλθουν από το Συμβούλιο για να λάβουμε ε, επικίνδυνε αποφάσεις. Εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να προστατεύσουν και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Για ένα λεπτό το λόγο και ο κύριος Πάντσα. Καλημέρα Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κλιματική αλλαγή υπολείπονται πάρα πολύ των προσδοκιών μας. Ω συνήθω χρησιμοποιήθηκαν ιδεολογικέ προσεγγίσεις που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Βερμπάνια, στο βόρειο Πιεμόντε, σε πολλέ περιοχέ τη Ιταλία, ότι έχουμε κατολιστήσει, πλημμύρε, κλειστού δρόμου, ακόμα και θανάτου. Δεν μπορούμε μέσω των φόρων να αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά επιτρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση να επέμβει, χωρίς να μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι στη φυλακή, χωρίς να θεωρείται ότι διαταράσσουν εσωτερική τάξη. Κάτι ακόμα. Το Ταμείο Λιλεγγύης, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτό το οποίο θεσπίστηκε και όχι για να καλύψουμε ζημίες που ενδεχομένω να προκύψουν από το Brexit. Α αφήσουμε άθικτο το Ταμείο αυτό προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να ταποκριθούμε στις ζημιές και τι φυσικές καταστροφές που πλήττουν όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Σίντσι τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τούσκ, κύριε Γιούγκερ, αγαπητοί συνάδελφοι, Βουρκώσατε και θα κρίσατε πριν από λίγο επειδή θέλει να αποχωρήσει το Ενωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας κάνει εντύπωση που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Εμάς μας είχαν πει ότι αυτή τη στιγμή στα μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαμε πλέον προβλήματα με τη διαφθορά. Δεν συμβαίνει όμω κάτι τέτοιο. Η χώρα μου, η Κροατία, εξακολουθεί και είναι μία από τι πιο διεφθαρμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το λένε επίσημε εκθέσει που δημοσιεύονται όλο και περισσότερο και εσεί αυτή τη στιγμή υποστηρίζετε ουσιαστικά το καθεστώ αυτό. Μπορεί για 10.000 ευρώ να εξαγοράσει κανείς τους δικαστές ή άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κροατία. Ξέρετε ότι πολύ συχνά στα πλαίσια των δικαστικών διαδικασιών στην Κροατία ρωτείται ένα ένοχο, ένα κατηγορούμενο, είστε ε, λοποδίτη, είστε κλέφτη. Αυτό απαντά δεν είμαι και κατευθείαν αθώνεται. Εμεί περιμέναμε ότι πραγματικά θα τοποθετούσετε πολύ πιο ψηλά τον πτήχη στην Κροατία, ότι θα επιβάλλετε υψηλότατα πρότυπα. Ανταυτού όμω εσεί δεχθήκατε τη στάση της κροατικής κυβέρνησης ε, σε διάφορα σκάνδαλα του παρελθόντος, αντί να επιβάλλεται τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα που υποτίθεται ότι έχουμε. Ο κ. Σόκολ, θα έχει μια, πράσινη μια μπλε κάρτα για σας. Δέχεστε, κ. Σέντσες. Μπλε κάρτα από τον κύριο Σόκολ. Θέλετε να απαντήσετε. Ωραία. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Σίντσιτς, δεν είναι η πρώτη φορά που εξαπατάτε και ψεύδεστε. Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί δεν θέλετε την, ε, το διορισμό Σουίτσα, ενώ η νομική επιτροπή έχει πει ότι είναι μια χαρά. Εξηγήστε μας. Για ποιο λόγο προσπαθείτε να ζημιώσετε την Κροατία. Go ahead. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ελπίζω να γνωρίζετε ε, τα ε, περί δωροδοκίας ε, βουλευτών είναι σε αποφάσεις ε, ποινικού δικαστηρίου της χώρας μας. Η Ευρώπη θέλει να εμπιστευτεί τα όργανα και τους θεσμούς της ε, Κροατίας που όμως είναι διεφθαρμένα. Είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκλεγεί επειδή ακριβώς ε, διαφωνούν με, τον, με αυτό που επικρατεί στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ε, Κύριο Στόμπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για το Brexit το καθοριστικό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποχωρήσουμε εμείς ή να υπαχθούμε στην εσωτερική ατζέντα, τις εσωτερικές προτεραιότητες του Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να καταλήξουμε γρήγορα σε μια συμφωνία όπως θέλει ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανυπόμονος, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί η παράταση ή, αν το αποφασίσει βέβαια το Βρετανικό Κοινοβούλιο, να περάσουμε σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα όπου θα αποφανθεί εκ νέου Βρετανικός λαός. Το πιο σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη συσπηρωμένη. Αυτή θα πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή μας και να αποφύγουμε βέβαια την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί συμφωνία. Το ιδανικό σενάριο βέβαια, η ιδανική έκβαση θα ήταν η, παρανομή, η παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αν είναι να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μια συμφωνία. Ο κύριο Μπενιφέ έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά απογοτευτικά τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να διαχειριστεί τις εξελίξεις που έχουμε παγκοσμίω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευτικό το ότι οι ηγέτες δεν κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά το πολιετές δομοσυνομικό πλαίσιο. Διαφωνούμε όλα με τις εισφορές, τους ιδίους πόρους, ακόμα και με τις περικοπές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν δεν ακολουθηθεί ο, ο ευκταίος οδικός χάρτης, να μειωθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτό πραγματικά θα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Είμαστε επίσης απλοί παρατηρητές της εισβολής της Τουρκίας στη Συρία. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επέμβει, να δημιουργήσει μία ζώνη απαγόρευσης των πτήσεων, να επιβάλλει κυρώσεις προκειμένου να μεταπιστεί η τουρκική κυβέρνηση και νομίζω ότι και στο ζήτημα αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πραγματικά να συμβάλλει προκειμένου να βγούμε από αυτό το καθεστώ παρατετημένη αδράνεια που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Μία ανακοίνωση για τις μπλε κάρτες. Θα σταματήσουμε με τις μπλε κάρτες γιατί έχουμε ακόμα 22 συναδέλφους εγγεγραμμένους στη διαδικασία Catch the Eye. Δεν μπορώ να δεχθώ από εδώ και πέρα μπλε κάρτε. Η κυρία Χαραντζόβα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Brexit ε, είναι η συζήτηση των ημερών. Θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για τις, ε, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τη διεύρυνση. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία έκαναν όλα όσα τους ζητήσαμε. Ε, έκαναν σημαντικές αλλαγές πληρώνοντας το πολιτικό κόστος. Τι είδους μήνυμα αποστέλουμε προς αυτούς σήμερα. Ε, για εκείνους οι οποίοι αντιτάχθηκαν στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνει ε, ξεκάθαρο ε, τι θα πρέπει να γίνει τώρα, τι δράσεις απαιτούνται. Θα πρέπει και θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να προβούν σε αυτές τις δράσεις με οικονομικά μέτρα η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία είναι ευρωπαϊκές ε, χώρες, ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό είναι καθήκον μας απέναντί τους να ξεκινήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος ε, Μπαρντέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε κάθε νέα διεθνή κρίση διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη διακρίνεται για την ανυμπόρια της. Ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν ομόφωνα την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, ε, δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε τον Ερντογκάν. Ε, παρά να τερματίσουμε τις άδειε εξαγωγής ε, όπλων στην Τουρκία. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, θα πρέπει να προβεί σε φορολόγηση των εξαγωγών της Τουρκίας. Ε, η Ρωσία δεν μπόρεσε να γίνει αντικείμενο τη ίδιας επίκαιες εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 19ο αιώνα λέγαμε για την Οθωμανική Αυτοκρατία ότι ήταν ο μεγάλο ασθενής της Ευρώπης. Αλλά σήμερα εμεί, οι Ευρωπαίοι είμαστε που είμαστε ασθενεί, ε, Ασθενεί από ένα ζωχισμό που μα υποχρεώνει να δίνουμε εκατομμύρια προ μια χώρα η οποία μας απειλεί να μα στείλει όλου του πρόσφυγε και συνεχίζουμε να τη θεωρούμε υποψήφια προς εισδοχή χώρα. Η κυρία Ντότζ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία ακόμα συμφωνία και μία ακόμα μεγάλη υποχώρηση και παράδοση από τον Μπόρις Τζόνσον. Στι 2 Οκτωβρίου <laughs> είχε πει ότι το, η Βρετανία, θα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να φύγει από, το, την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο. Ε, η, όμως ε, ε, οι επιχειρήσει στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, θα πληρώνουν φόρου κατά βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμόζουν του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα χτε επιβεβαιώθηκε ότι τα αγαθά τα οποία θα έρχονται από τη Βόρεια Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα περνάνε από τελωνιακέ διαδικασίε με κόστο 65 ε, περίπου λίρες ανατελωνιακή αποσαφήνιση. Ε, δεδομένου ότι ε, τεράστιος όγκος εμπορίου γίνεται μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας, το κόστος είναι τεράστιο αν η Βόρεια Ιρλανδία αποκλει... απο... από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας ε... φημισμένος ε, οικονομολόγος ε, είπε μάλιστα ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι παρατηρήτρια σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπόρις Τζόνσον υπέγραψε κάτι το οποίο κανεί ε, Βρετανός Πρωθυπουργός δεν θα έχει υπογράψει παλιότερα. Ευχαριστώ. Ο κ. Νίτερ Μάγερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για το Brexit. Θέλω να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ίδιο. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Τούσκ και τον κύριο Γιούνκερ για την αφοσίωσή τους, για τις προσπάθειές τους ε, και στο τελευταίο Συμβούλιο αλλά και στα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώ όμως μερικές φορές η απροσύλωση και οι προσπάθειες δεν είναι αρκετές. Το θέμα είναι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί συνεργασία και να γίνει κοινή προσπάθεια για το μέλλον. Ή είναι το όργανο στο οποίο λαμβάνουν χώρα πολιτικά παιχνίδια μόνο. Έχω την εντύπωση ότι τελευταίο, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο υπερτέρησε του πρώτου. Ελπίζω να είναι η εξαίρεση, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Mr. Schieder, for one minute. Ο κ. Σίντερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε το Brexit ε, μεταγράφεται σε μια τέρμονη ιστορία. Είναι ο τρίτος ε, Βρετανός Πρωθυπουργό που ασχολείται με το θέμα αυτό και η κατάσταση επιδενώνεται συνεχώς. Η αποτυχία του Brexit είναι αποτέλεσμα του διχασμού των Τόρις. Είναι το αποτέλεσμα του, του εγωισμού του Βρετανού Πρωθυπουργού Boris Τζόνσον και πρόκειται για ένα εγωιστικό παιχνίδι βάρος των ε, πολιτών, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ε, χρειάζεται το Brexit, ε, χρειάζεται και μια λογική συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το Brexit συνεπάγεται μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, μείωση της προστασίας των καταναλωτών, λιγότερους πόρους και συνεπώς είναι μια κακή ιδέα. Ε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας να διαπράξουμε ένα σφάλμα. Αλλά εμεί οι ίδιοι δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα σφάλμα. Γι' αυτό θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει για τη συμφωνία μόνο εφόσον ε, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο με τα, με τα δύο του σώματα λάβει αυτή την απόφαση και μετά είναι η δική μας σειρά. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κούτσουκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν πολύ σημαντικό γιατί έγιναν προσπάθειες να ξεπεραστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Βόρεια Συρία. Επίσης έγιναν προσπάθειες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια, να επιταχθεί μια συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο το Brexit επίσης. Η Μεγάλη Βρετανία θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπόρις Τζόνσον ήθελε να γίνει αυτό τέλος Οκτωβρίου, αλλά δεν είχε ξεκάθαρο στόχο. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την παράταση του Brexit, γιατί ε, είδαμε τι επιθυμούν οι πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορώ παρά να αναφέρω το ιστορικό σφάλμα το οποίο έγινε όσον αφορά την ε, ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Κάθε αναβολή της ε, ενταξικής διαδικασίας συνιστά σφάλμα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση της περιοχής και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χώρες αυτές. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Η κυρία Γκάντσα έχει το λόγο. Από τι φαίνεται απουσιάζει όμως ο κύριος Χριστοφόρου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω πραγματικά τις πολύ σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να λάβει μέτρα ενάντια στην επιθετική επεκτατική δραστηριότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τούσκ που δια τη παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτά τα πέντε χρόνια μαζί και με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. ζαν κλοντ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναβάθμισαν με το έργο τους και την αποστολή τους το κύρος και την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ένωσης. η τουρκία εισέβαλε στη συρία κατά τον ίδιο και ανάλογον τρόπο ανενόχλητο που εισέβαλε πριν 45 χρόνια στην κύπρο μας και άφησε πίσω τη όλεθρο και καταστροφή. από τούτο εδώ το βήμα προειδοποίησα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει εδώ και τώρα να αναχαιτήσουμε την επεκτατική και επιθετική πολιτική της Τουρκίας για να μην είναι αργά. και για να μην είναι αργά πιστεύω ότι οφείλουμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του αγαπητού φίλου ηγέτη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο Μάφρε Βέμπερ, που ξεκάθαρα είπε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να απολαμβάνει την Τελωνιακή Ένωση, την εσωτερική αγορά και να στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εισβάλλει σε χώρε όπω τη Συρία αλλά και παραβιάζει αρχέ και δικαιώματα. Οφείλουμε όλοι αυτή τη στιγμή να τοποθετούμε και να υιοθετήσουμε την πρόταση του Μάφρε Βέμπερ για να υπάρξουν οικονομικέ συνέπειε ενάντια στην Τουρκία. Μόνο έτσι η Τουρκία θα καταλάβει και θα κατανοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση αρχών και αξιών και ουσιαστικά οφείλουν όλοι να την αναγνωρίζουν και να τη σέβονται. αλλά ταυτόχρονα τελειώνουν τα κυρία πρόεδρε μόνο έτσι η ευρωπαϊκή ένωση θα αποδειχθεί επιτέλου ότι είναι ηγέτιδα δύναμη και θα γίνει σεβαστή και από εχθρού και φίλου. ευχαριστώ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας δεν νομίζω ότι τα πράγματα κινήθηκαν ως συνήθως γιατί είχαμε πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία επισκίασαν την όλη συζήτηση όπως για παράδειγμα το Brexit και αυτό φάνηκε τελικά από το, τα συμπεράσματα ιδίω για τον ε, για την υπόθεση της Συρίας δεν έχουν πολλές ουσιαστικές παρατηρήσεις, το ίδιο και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. και λυπάμαι πάρα πολύ που μολονότι μιλήσαμε τόσο εκτενώς για το Brexit δεν καλύψαμε παρκώς τη μη έναρξη συνταξικών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ζήτημα το οποίο πραγματικά βάλει καλά τις ίδιες τις αξιοπιστίες μας και τις παρουσίες μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκες διεθνές προκλήσεις στην όλη αυτή περιοχή και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σαφώ θα πρέπει στα πλαίσια του Brexit να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τη στάση των Βρετανών πολιτικών. Α μην ξεχνάμε όμω ότι από εμά ε, εξαρτώνται όλε αυτέ οι κυβερνήσει οι οποίε κάνουν μεταρρυθμίσει, όπω υποψήφιε χώρε. Ο κύριο Ρανχέλ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να φανταστούμε χωρίς τον πρόεδρο Γιούγκερ μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα τελευταία χρόνια. Και σας ευχαριστώ πραγματικά και σας τιμώ όχι μόνο για την πολιτική σας δραστηριότητα, αλλά γιατί πραγματικά ήσασταν ένας αληθινός ουμανιστής και ένας πραγματικός Ευρωπαίος. Και να σας πω ότι ε, το ακόλουθο δόγμα του Μονσκέ πραγματικά συνοψίζει τα όσα θέλω να πω. Αν πραγματικά υπήρχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο για την Ευρώπη και θα ήταν αρνητικό για την ανθρωπότητα, αυτό θα ήταν πραγματικά ένα έγκλημα. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο συνοψίζετε πραγματικά η συλλογιστική σας και η δράση σας. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτον, συμφωνώ πλήρως με τις θέσεις σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το, με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί για το βρετανικό λαό, διατηρώντας όμως την προστασία του ευρωπαϊκού οράματος. Ε, προασπίζοντας την Ευρώπη, προασπίζουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερον, προερχόμενος από το Far West της Ευρώπης, να σας πω δύο λόγια για τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι ντροπή που δεν είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει ένταξη με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Μα χρειάζονται τόσο όσο και εμεί οι ακροδυτικέ χώρε τη Ευρώπη ε, χρειαζόμαστε την Ευρώπη στο παρελθόν. Thank you. For one minute, Mr. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό ο λόγος στον κύριο Μορένο Σάντσες. Ζων Κλοντ Μισελ, έχω ένα μόνο λεπτό, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κυρίες και κύριοι, το Brexit μας διατηρεί σε μια απόλυτη αβεβαιότητα. Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων εξακολουθεί να επικρατεί χάος και αβεβαιότητα. Καλύτερο να αναβάλουμε την αποχώρηση παρά να δεχτούμε ένα σκληρό Brexit. Χρειαζόμαστε όμω ταυτόχρονα και ένα φιλόδοξο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα υπερβαίνει κατά πολύ το 1% του ΑΕΠ. Ορισμένοι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων το είπαν, μεταξύ αυτών και ο δικό μου Πρωθυπουργό. Επίση έχουμε το, την πρόκληση τη κλιματική αλλαγή, τη ε, ψηφιακής ατζέντα και τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε χρήματα γι' αυτό. Επίση χρειαζόμαστε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την αργία των νέων, την μακροχρόνια ενεργεία κλπ. Και επίση θα πρέπει να ενισχύσουμε την ΚΑΠ, την περιφερειακή συνοχή και την οικονομική κοινωνική συνοχή. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε η ύπεθρο να ερημώνει και να μεγαλώνει διαφορά ανάμεσα στην ύπεθρο και τις πόλεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Σκέλη, ένα λεπτό. Ε, η 31η Οκτωβρίου είναι πολύ κοντά. Και ταυτόχρονα έχουμε και το Halloween, ε, το καρναβάλι, ε, τα φαντάσματα και άλλα τρομακτικά πράγματα. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αφιερώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε σωστά με την ε, Συμφωνία Αποχώρηση. Ήδη έχουν περάσει τρία χρόνια. Γιατί να βιαστούμε. Α δώσουμε στον εαυτό μα μερικού μήνε ακόμα. Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρηση είναι σίγουρα καλύτερη από ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Και θέλω να συγχαρώ και τον ε, Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και τον Μπόρις Τζόνσον και τον Μισελ Μπαρνιέ για τι προσπάθειε τους. Α δώσουμε χρόνο στον εαυτό μα να τα καταφέρουμε σωστά. Επίσης, τελικά, θέλω, και στο τέλο, θέλω και εγώ να συγχαρώ τον πρόεδρο τη Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, ήταν εξαιρετική θητεία του. Έδειξε οι ικανότητε και η Ευρώπη θα του χρωστά για πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι, 22 αιτήματα για catch ε, the eye. Θα, πάρω, ε, θα δεχθώ μόνο 7. Ο κύριος Κίρτσος πρώτος. Με ανησυχεί ότι υπάρχει μια κακοφωνία μεταξύ Μέρκελ και Μακρόν, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Σε πολλά ζητήματα βρίσκονται αντίθετοι από τη χρηματοδότηση της ευρωζώνης από τη διεύρυνση στα δυτικά βαλκάνια από την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής από τη σχέση με τη ρωσία. επομένως θα ήθελα να ξεπεραστεί αυτή η κακοφωνία γιατί πιστεύω ότι με μια καλύτερη γαλλογερμανική συνεργασία θα αποκτήσουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Γιούνκερ για ό,τι έκανε για την πατρίδα μου την Ελλάδα. Όλοι τον ευχαριστούμε στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση διότι ο Γιούγκερ αγαπάει τους έλληνες μας αγαπάει όλους με τις γνωστές αδυναμίες και τις ελλείψεις μας. άλλωστε αυτή είναι η πραγματική έννοια της αγάπης να είναι ανιδιοτελής. τον ευχαριστούμε πολύ για όσα έκανε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βόρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίζει παιχνίδια με όλες μας. Ήταν ευτυχής να ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα του κυρίου Μπόρις Τζόνσον για το Brexit, αλλά όχι να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το Συμβούλιο ήταν ε, πρόθυμο σε σχέση με το Brexit αλλά δεν ήταν εξίσου πρόθυμο να δείξει υπομονή με τους, ε, να τιμήσει τη συμφωνία με τους γείτονές μας και αυτό συνιστά ένα σφάλμα όσον αφορά το Ενωμένο Βασίλειο τι είδου ε, διεθνή συμφωνία θα έπρεπε να επισπεύσουμε χωρίς μια σωστή αξιολόγηση το Συμβούλιο θέλει να μετακυλήσει την απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να μας επιτρέψει ικανό χρονικό διάστημα για να το εξετάσουμε. Το Brexit δεν θα γίνει ως διαμαγείας. Εάν αν περάσει το Brexit ε, θα έχουμε... Ε, τώρα θα ξεκινήσουν οι μεγάλες δυσκολίες. Ο κύριος Σάνσιπ, ο έχει το λόγο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Ζαν Κλόντ Τόναλτ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Ζαν Κλόντ για την πολύ καλή ηγεσία που έδειξε. Αλλά για το Brexit μετά το δημοψήφισμα είχαμε πολύ ισχυρέ δηλώσεις από το Λονδίνο. Μας λέγανε το Brexit σημαίνει Brexit. Έξοδος σημαίνει έξοδος. Καλύτερα να μην έχουμε συμφωνία από το να έχουμε μια κακή συμφωνία. Ως Επίτροπος για τα ψηφιακά ζητήματα κατάφερα να ασχοληθώ με δύσκολα ζητήματα κατάργηση των τελών περιαγωγή, για παράδειγμα. Τι θα γίνει όμω με τα τέλη περιαγωγή μετά τον Brexit, θα εξαρτηθεί από τι διαπραγματεύσει μεταξύ του Μένου Βασιλείου και των 27 κρατών μελών. Καταφέραμε να έχουμε ένα κανονισμό προστασία τη ιδιωτική ζωή των πολιτών. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την ελεύθερη ε, διάδοση και διαβίβαση των δεδομένων για τι επιχειρήσει μα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το Μένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά την παροχή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του cloud. Τι θα γίνει όμως με την ροή των δεδομένων μετά το Brexit. Πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις. Συγγνώμη, ολοκληρώθηκε το ένα λεπτό, κύριο Άνσιπ, και είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο τώρα έχει ο, επόμενο ομιλητής, κυρία Τσάνς, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σε ευχαριστήσω όλου για την υπομονή σα με τον εφιάλτη του Brexit. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την εξέλιξη κατάσταση και εγώ θεωρώ ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια και συμφωνώ μαζί σα. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει τώρα να επισπεύσουμε τεχνικό πώ τα πράγματα και εγώ συμμετείχα στι πορείε που έλαβαν χώρα το Σάββατο στο Λονδίνο ζητώντα δεύτερο δημοψήφισμα. Θα είδατε τι εικόνε με πραγματική θάλασσα ανθρώπων που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Αυτή είναι η βούληση του λαού και άλλαξε από το 2016 στο παρελθόν, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, στο 74% των περιπτώσεων, είδαμε ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι υπέρ τη παραμονή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλα αυτά έχουμε έναν νέο Πρωθυπουργό, ο οποίο έχει χάσει κάθε ψηφοφορία που έχει γίνει στη Βουλή των Κοινοτήτων, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν, και τώρα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον βγάλει από το χαντάκι στο οποίο ο ίδιο μπήκε από μόνο του. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση στο Westminster. Γνωρίζουμε όμω ότι ο στόχο των υπερμάχων του Brexit είναι να απολέσουν την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε εμείς σε καμία περίπτωση να υποστηρίξουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ο κύριος θα έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Has been a good customer and friend of the European Union and its member states. In the 20 years to 2018, the EU enjoyed a total trade surplus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 Ο κύριος Μπόκοβιτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τούσκα γιατί ήταν η φωνή της λογικής τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα προορατική στάση του κυρίου Γιούνκερ για τα καταπληκτικά αποτελέσματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit και αναφέρομαι στον κύριο Μπαρνιέ. Κατάγομαι από τη Σλοβενία. Και μας συντάραξε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ξεκινήσει ενταξιακέ διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Προερχόμαστε από μια περιοχή που γνωρίζουμε ότι η ειρήνη δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Ξέρω ότι πολλές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν ακόμα στις δύο αυτές χώρες, αλλά δυστυχώς τα μηνύματα αυτά τα οποία στέλνει τώρα το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσοι εξημών γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την περιοχή της Ευρώπης, όσοι από εσά επισκέπτεστε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χώρε αυτέ βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ την Επίτροπο Χάν για τα πολύ θετικά αποτελέσματά του στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή θα αλλάξει η ισορροπία στην όλη περιφέρεια εξαιτία τη πολύ αρνητική αυτή απόφαση. Gracias, señora presidenta. Λόπεθ Αγγιλάρ. Κύριε Γιούνκερ, πρόεδρε Γιούνκερ, θέλω κι εγώ να, γνωρίσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ε, βρισκόμασταν στην χειρότερη κρίση μας ε, με επικεφαλή στο Brexit. Το καλό νέο μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας σας ήταν ότι τι ε, διατρήσαμε την ενότητά μα. Ε, και ε, αυτό οφείλεται και στον κύριο Μπαρνιέ, γιατί εξασφαλίζουμε και την αμοιβαιότητα. Δηλαδή, εμεί θα φερθούμε στο, στου Βρετανού πολίτε εδώ στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο αυτοί θα φερθούν στου δικού μα πολίτε στην δική του επικράτεια. Ε, όμως, ε, τα ιαλουχία των γεγονότων μας οδηγεί σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία και τα οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, ειδικά οι πολιτικές επιπτώσεις, διότι οι εθνικιστές έχουν προβεί σε μια εκστρατεία δηλητηρίασης του πολιτικού βίου με ψέματα. Θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη, αλλά για αυτή τη μάχη χρειαζόμαστε πόρους και με το 1% του ΑΕΠ δεν θα το καταφέρουμε. υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στα λόγια και, στα, και στις πράξεις και θα πρέπει να την ξεπεράσουμε. Δεν είναι δυνατόν άλλα να υποσχόμαστε και άλλα, με άλλα να συμμορφόμαστε. Συμμορφωνόμαστε τελικά. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Παρνιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, με την άδεια του κυρίου Τους και του κυρίου Γιούγκερ θα ήθελα να πω κάποια λόγια για να απαντήσω σε όσους ε, ε, μίλησαν σε σχέση με αυτό το δύσκολο θέμα του Brexit. Τον κύριο Βέιμπερ, την κυρία Γκαρσία Περές, τον Φίλιπ Λάμπερτς και όλους πόσους ε, τα τελευταία τους τελευταίους μήνες με στήριξαν την εμπιστοσύνη τους. Όπως είπε ο κύριος Τούς και ο κύριος Γιούγκερ, έχουμε μεγάλο σεβασμό για το σώμα σας. Έχουμε πάντοτε ε, και είναι το δικό σα κοινοβούλιο αυτό το οποίο θα έχει την τελευταία λέξη. Άρα είναι φυσιολογικό το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει τώρα τις ευθύνες του και να δεσμευθεί πρώτο στη βάση της συμφωνίας που έχουμε διαπραγματευθεί με την Βρετανική κυβέρνηση και όχι ενάντια στη βούληση της Βρετανικής κυβέρνησης ή ερήμην της Βρετανικής κυβέρνησης προκειμένου να πετύχουμε το ε, ένα συντεταγμένο Brexit. Και το επαναλαμβάνω, εάν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί ένα συντεταγμένο Brexit, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από μια άτακτη έξοδο, η συμφωνία αυτή είναι η μόνη δυνατή. Και μας φαίνεται θεμητό ε, το δικό σας σώμα να δώσει πριν δώσει την συγκατάθεσή του να γνωρίζει χωρίς αμφισημίες τι επιθυμεί, τι αποφασίζει, τι το Ηνωμένο Βασίλειο για το μέλλον του. Άρα βρισκόμαστε σε μια σημαντική ε, φάση αυτής της μακράς διαδικασίας και ε, είχα την ευκαιρία να το πω και στον κύριο Τούσκ και στο επιτελείο του καθώς και στον κύριο Γιούγκερ και στον πρόεδρο του, και στον κύριο Βέρχοφ Στάτ, ε, τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του. Ε, η αποστολή που μου ανατέθηκε, που από τον κύριο Γιούνκερ, είναι να εργαστώ για να οργανώσω μία συνδεταγμένη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας και όχι κάτι διαφορετικό. Και είναι αυτό το οποίο, στο οποίο καταλήξαμε. Ωστόσο ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή γιατί πρόκειται για μια αρνητική διαπραγμάτευση στην ουσία, όπου όλοι θα βγουν ε, χαμένοι. Ούτε ο κύριος ε, Φαράτζ δεν ήταν ε, ικανός να μου αποδείξει την προσθέμενη αξία του Brexit. Άρα λοιπόν έπρεπε να κάνουμε μια αρνητική διαπραγμάτευση, λαμβάνοντας τη σοβαρά, ούτως ώστε να σεβαστούμε τη Βρετανική απόφαση, έστω και αν ε, λυπούμαστε για αυτήν. Ε, εργαστήκαμε λοιπόν με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα ε, προσπαθώντας να εξεύρουμε λειτουργικές και νομικά αποδεκτές λύσεις προκειμένου να επιλύσουμε το κάθε πρόβλημα που θέτει το Brexit. Ε, και αυτό από όλες τις πλευρές και για όλο τον κόσμο. Σεβαστήκαμε τους εταίρους μας, τους Βρετανούς, γιατί κύριοι βουλευτές έχουμε σεβασμό για το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα και αισθήματα θαυμασμού. Εργαστήκαμε λοιπόν χωρίς ε, να επηρεαστούμε από τις ε, ενδοβρετανικές ε, ταραχές και αντιπαραθέσεις. Γιατί υπήρξαν πολλά προβλήματα που θέτει το Brexit. Εργαστήκαμε λοιπόν με την προοπτική αυτής της διαπραγμάτευσης. Αλλά ωστόσο το Brexit δεν είναι ένα πεπρωμένο, δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Ε, αντιμετωπίσαμε τη διαπραγμάτευση αυτή υπό το πρίσμα της ειρήνης στην Ιρλανδία, γιατί καθημερινά υπήρξε αυτό το επιτακτικό αίτημα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διατηρήσουμε αυτή την ε, τροτή ειρήνη, την ευάλωτη ειρήνη στην Ιρλανδία. Επίσης όσον αφορά τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς η οποία είναι κάτι παραπάνω από μια χώρα ελεύθερων αλλαγών αλλά είναι ένας χώρος κοινής διαβίωσης και συνύπαρξης και θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί. Επίσης ε, λάβαμε υπόψη μας τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ε, πολιτών ε, υπάρχουν 3,5 Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι διαβιούν σε Αρμένο Βασίλειο και αντιστρόφως υπάρχουν πολλοί ε, πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας που ζουν στην Ευρώπη και θα πρέπει να μερμηνήσουμε για αυτούς. Εάν η συμφωνία αυτή ψηφιστεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και από εσά, τα 4,5 εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και για τις οικογένειές τους. Είναι, αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή και θέλουμε να το επαληθεύσουμε. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την πίεση ούτως ώστε οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρηθούν. Επίση, ε, κάναμε αυτή την διαπραγμάτευση εφόσον το Brexit δεν είναι σαν το τέλος τη ιστορία. Ε, να δούμε αυτό το οποίο θα οικοδομήσουμε από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία. Η, η Μεγάλη Βρετανία θα εγκαταλείψει πάνω από 600 ε, διεθνείς συμβάσεις, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Θα παραμείνουν οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας, οι εταίροι μας. Άρα θα πρέπει να προβούμε και μια, σε μια διαδικασία να Ανοικοδόμηση, αν θέλετε. Ο κ. Φάραντς δεν ε, ε, παρίσταται εδώ γιατί λέει ότι η συμφωνία αυτή θα ανοίξει ε, ένα διάστημα τριών ετών νέων διαπραγματεύσεων. Μα φυσικά είναι η απάντησή μας. Θα πρέπει ε, να ξαναφτιάξουμε όλα αυτά τα οποία ξυλώσαμε μέσω του Brexit. Θα πρέπει να φτιάξουμε ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες σεβόμενοι τους κανόνες παιχνιδιού για να αποφύγουμε τους κινδύνους ενός ε, οικονομικού, κοινωνικού, υπερεβαλλοντικού dumping ε, ε, διατηρώντας τις συνεργασίες σε πανεπιστημιακό επίπεδο στο πλαίσιο του Εράσμους, στο πλαίσιο της ε, συνεργασίας μεταξύ των, αστυνομιών, των, των αστυνομικών αρχών των υπηρεσιών και λοιπά και λοιπά, της δικαστικής συνεργασίας. Όλα αυτά τα οποία ξυλώνονται λοιπόν θα πρέπει να τα επανοικοδομήσουμε με τη Μεγάλη Βρετανία θα ήθελα να καταλήξω αναφερόμενο στα όσο είπε ο κ. Βανόρντεν, ο οποίο είπε ότι υπάρχει ένα δίδαγμα το οποίο θα πρέπει να αντλήσουμε από το Brexit. Οι συνέπειε του Brexit, οι οποίε θα είναι αναρρύθμιτε και οι οποίε συχνά υποτιμήθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία και οι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί 50 ε, τόσοι, 100 ε, ε, ε, ψήφισαν, καταψήφισαν την Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχει ένα μάθημα, ένα δίδαγμα το οποίο θα πρέπει να αντλήσουμε. Κάτι το οποίο συχνά λησμόνησε ο κύριος φάρατ ότι θα πρέπει να πει κανείς την αλήθεια στους πολίτες πριν πάνε στις κάλπες. Αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε, που φέρουμε έναντι των πολιτών. Αλλά πίσω από την ψηφοφορία για τον Brexit υπάρχει και ένας κοινωνικός θυμός που εκφράστηκε γιατί η Ευρώπη πολλές φορές ε, δεν ε, σέβεται αρκετά τα συμφέροντα των πολιτών της στο πλαίσιο της των οικονομικών εξελίξεων. Ε, ελπίζω ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν θα δώσει προτεραιότητα στο νέο αυτό πολιτικό ευρωπαϊκό θεματολόγιο αλλά θα ήθελα να πω ότι ήταν και δέσμευση του κυρίου Γιούγκερ ε, και των επιτρόπων του και του σώματος των επιτρόπων, τους οποίους θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Ε, πέραν των ορίων του Brexit θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική δέσμευση για ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπαρνιέ. Τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Ντόναλτ Τούσκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα τα θετικά λόγια που είπατε για το πρόσωπό μου. Άξιζε να περιμένω πέντε χρόνια για να ακούσω τα καλά αυτά λόγια. Σας ευχαριστώ επίσης για την υπεύθυνη στάση που δείξατε απέναντι στο Brexit και για το ζήτημα της παράτασης. Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά δείξατε μια στάση αξιοπρέπειας. Μετά τα όσα άκουσα σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω αναμφίβολα ότι θα πρέπει να δεχθούμε και να εξετάσουμε με απόλυτη σοβαρότητα το αίτημα των Βρετανών για παράταση. Σας ευχαριστώ πολύ και σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσουμε για τη διαθεσιμότητά σας πάντα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες αυτές τις ζητήσεις που κάναμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ προφανώς για τη δέσμευση και την προσήλωσή σας. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Cominciamo. Ξαναρχίζουμε. Καθίστε παρακαλώ. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητέ Πρόεδρε Γιούνκερ, Σήμερα είμαστε εδώ για τον απολογισμό της ε, Επιτροπής σας. Ευχαριστώ τους επιτρόπους που είναι παρόντες εδώ στην Ολομέλεια και πριν ε, σας δώσω το λόγο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας ε, στην υπηρεσία της Ευρώπης. Μια δέσμευση η οποία δεν ξεκίνησε όταν εκλεγήκατε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως κύριος υποψήφιος, επικεφαλής ε, του ψηφοδελτίου, αλλά ήταν στη διάρκεια όλου του επαγγελματικού βίου. Στη διάρκεια τη Προεδρία σα αποδείξατε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να απομονώνει, αλλά να ενώνει στις διαπραγματεύσει για τον Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω τη αναζήτηση μια ευρωπαϊκή απάντηση ε, στο πλαίσιο τη μεταναστευτική πολιτική και τη υποδοχή των προσφύγων, στην καταπολέμηση του λαϊκισμού, στο σχέδιο Juncker, αλλά και στην εμβάνθηση τη ΟΝΕ, και την ε, παραμονή της Ελλάδος ε, στην Ευρωζώνη οι προκλήσεις ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλες και παρά τις ε, διάσταση απόψεως, ε, τις συζητήσεις που αποτελούν και ένδειξο της ζωντάνιας της δημοκρατίας, πάντα μπορούσατε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια πιο δίκαιη, πιο ενωμένη, πιο βιώσιμη και πιο κοντινή στους πολίτες Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε επίσης και για την συνεργασία και για την προσοχή που δείξατε ανέκαθεν για το Κοινοβουλίο μας. Έχετε το λόγο, Πρόεδρε Γιούνκερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Πέντε χρόνια ακριβώς, μέρα με τη μέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε την εμπιστοσύνη του στην Επιτροπή μου και ποτέ δεν με διαψεύσατε, ποτέ δεν με αμφισβητήσατε. Ορισμένες φορές ήταν δύσκολες οι σχέσεις μας, ε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πάντα ήταν ευγενείς. Ε, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, ε, διότι το να διαθέτω την εμπιστοσύνη αυτού του ημικυκλίου, το να μπορέσω να βασιστώ στην εμπιστοσύνη των ερετών ε, της Ευρώπης, ε, αντανακλά την ευρωπαϊκή δημοκρατία και για τον καθένα από εμά το να εκλαμβάνει αυτή την εμπιστοσύνη είναι μια διαρκή τιμή. Βλέπω εδώ πολλέ οικίες φυσιογνωμίες, ε, πολλού οι οποίοι έγιναν φίλοι, όχι μόνο ε, εντό των θεσμικών οργάνων, αλλά φίλοι διαβίου και γι' αυτό θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ βάθου καρδία, όπω ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Τούσκ. είμαστε δίδυμοι αλλά ακόμα και οι δίδυμοι ορισμένες φορές μπορεί να διαφωνούν. Είχαμε όμως την ξυπνάδα να ε, κρύβουμε αυτές τις διαφωνίες μας και για σας ίσως να αποτελεί έκπληξη ε, το γεγονός ότι είχαμε και κάποιες διαφωνίες αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντόναλτ ε, για την βοήθειά του για έναν φίλο ο οποίος θα παραμείνει φίλος και είναι τιμή να τον έχω φίλο μου ε, οι, αμυσ... οι φιλίες ορισμένες φορές στην πολιτικό βίο είναι σπάνιες ιδιαίτερα εντός της ίδιας πολιτικής οικογένειας είναι πολύ πιο σπάνιες και με τον Ντόναλτ όμως ε, δεν θα χωρίς μάλλον τον Ντόναλτ δεν θα μπορούσα να ίσα κάνει αυτά που έκανα και επειδή είναι η τελευταία φορά που απευθύνω τον λόγο εδώ στο ημικύκλιο, θα ήθελα να ευχηθώ και καλή τύχη στην κυρία Φόντερ Λάιεν, που είναι ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η οποία χρειάζεται και την ενθάρρυνσή μας ε, και κάθε ευχή είναι ευπρόσδεκτη. Της εύχομαι λοιπόν ούριο άνεμο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιτρόπους μου. Διότι χωρίς αυτούς πάλι δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα. Είναι άνδρες και γυναίκες οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συλλογικά είναι άνθρωποι που τους άξιζε η Ευρώπη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστή σε διάφορες γλώσσες ο Πρόεδρος. Από τότε που ανέλαβα καθέκοντα το 2014, η Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη. Υπήρχαν ρήξει ε, στην αλληλεγγύη, πολλαπλές και η Ευρώπη το 2014 δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, γι' αυτό και μίλησε και για την Κομισιόν της τελευταίας ευκαιρίας. Δεν θα είχα μιλήσει όμως ε, για την Κομισιόν, αλλά για μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπηρεσία της Ευρώπης που έχει κάποια βλάβη, διότι το 2014 βρισκόμασταν σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης και γι' αυτό ακριβώς όλοι είχαμε αναλάβει να ε, εκμεταλλευτούμε αυτή την τελευταία ευκαιρία η οποία είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Ευρώπης μαζί με τους ε, συναδέλφους μου προσπάθησα να στήσω μια πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα η Επιτροπή να είναι ερετή. Ε, πέραν ε, του Βρετανού Επιτρόπου. Είχα δύο Βρετανούς Επιτρόπους, τον έναν πιο εξαιρετικό από τον άλλον, αλλά όλοι οι Επίτροποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήθελα η Επίτροπη να είναι οικία πρόσωπα στις χώρες τους αλλά και στην Ευρώπη και τους είχα προσκαλέσει να μην σταματήσουν στις Βρυξέλλες, να μην κλειστούν στον Περλεμό, αλλά να κυκλοφορούν και να εξηγούν, να συνομιλούν με τους υπόλοιπους ερετούς και φυσικά και με την κοινή γνώμη και με τους πολίτες. Στη διάρκεια αυτών των πέντε ετών διοργανώσαμε 195 διαλόγους με τους πολίτες ε, και ε, οι επίτροποι ε, επισκέφτηκαν 911 φορές τα εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερικά κοινοβούλια. Πέραν αυτού στην αρχή της ηττίας σας είχα υποσχεθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχε σταθεί μόνο στα βασικά. Θέλαμε να είμαι big on big και να προχωρήσουμε και σε μεγάλα θέματα. Θέλαμε να ε, θέσουμε ένα τέλος σε αυτό τον πληθωρισμό που είχαμε στην νομοθεσία, η οποία χαρακτήριζε μέχρι τώρα τη δράση, μέχρι τότε μάλλον, τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε 84% λιγότερες νομοθετικές προτάσεις σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή. Ε, αποσύραμε 142 νομοθετικές προτάσεις και εξυγχρονίσαμε 162 ε, κείμενες ε, νομοθετικές ε, πράξεις. Ποιος λοιπόν άλλος έκανε αυτά που είχε υποσχεθεί. Βέβαια υπήρξαν διάφορες φωνές οι οποίες ε, ήταν επικριτικές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλεγαν ότι ε, ασχολούμαστε με τα πάντα και ότι προδικάζουμε τα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ε, άλλαξαν τα πάντα, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ ενώπιόν σας Και εγώ είχα τρία πράγματα που ήθελα να αποτελούν ε, τις επιταγές της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάπτυξη, επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης. Και είμαστε στο πέμπτο ε, συνολικό τρίμηνο ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχουμε δημιουργήσει 14.000 ε, ε, θέσεις εργασίας. Έχουμε ε, την πιο μεγάλη ανάπτυξη. 241.000 ευρώ, εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι σε θέσεις απασχόλησης και αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα καλύτερα ποσοστά. Το σχέδιο Juncker οδήγησε και σε επενδύσεις και είχαμε 432 δισεκατομμύρια. Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι πίστευαν ότι το σχέδιο Juncker θα είναι αποτυχία ε, και μιλούσαν για την επιτυχία του Juncker, τώρα που είναι επιτυχία ε, αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκό μέτωπο επενδύσεων. Έτσι είναι η ιστορία. Ένα εκατομμύριο θέσεις εργασία δημιουργήθηκαν χάρη στο σχέδιο Juncker. Και Κάναμε και μια νέα ανάγνωση για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, δίνοντας ευελιξία σε κάποιες από τις διατάξεις του και το κάναμε παρά τη θέληση πολλών. Ε, πολλών κρατών μελών που ποτέ επισήμως ε, δεν ενέκριναν τις γραμμές της ευελιξίας τις οποίες χρησιμοποίησαμε για να εμπλουτίσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά ε, τα ελλείμματα από το 6,6% πέρασαν στο 0,7%. Αυτή η ευελιξία λοιπόν, την οποία ε, σκεφτήκαμε και ήταν αρκετά έξυπνη για το Σύμφωνο Σταθερότητας, μας βοήθησε να ανταποκριθούμε στο παρόν, γιατί η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα είχαν ζητήσει να δράσουμε ε, για να τις βοηθήσουμε. Αγαπητοί φίλοι, ε, είχα και κάποιες απογοητεύσεις ε, στην θητεία μου. Απογοητεύσεις διότι δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε τα θέματα της επανένωσης της Κύπρου. Εκεί χάσαμε χρόνο και δεν μπορέσαμε να συνάψουμε μια συμφωνία με την Ελβετία. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε, οι οποίες ήταν πολυάριθμες και εντατικές. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Όχι ελήψη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χάρη ή ε, λόγω ελλείψεως προσπαθειών των κρατών μελών. Αν δεν ολοκληρώσουμε όμως την Τραπεζική Ένωση όπως πρέπει, κάνοντας την Οικονομική Νομισματική Ένωση, μια Τραπεζική Ένωση που να εκπροσωπεί ε, την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους κλειδονισμούς. Είτε οι κλειδονισμοί οικονομικοί είναι εσωτερικοί ή προέρχονται έξωθεν. Είναι ανάμεσα αυτά πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων. Χωρίς εγγύσει καταθέσεων δεν υπάρχει τραπεζική ένωση και χωρίς εγγύσει καταθέσεων δεν υπάρχει τραπεζική ένωση και χωρίς τραπεζική ένωση τέλεια δεν έχουμε πλέον οικονομική και νομισματική ένωση. Πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις παρά την πολλαπλή ε, κρίση συγγνώμη, των τελευταίων πέντε ετών, τη δική μας κρίση, είχαμε και επιτυχίες. Δεν τολμώ να πω επιτυχίε. δεν θέλω να δείξουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι στου παθιέ μα, παρά το ότι θα ήθελα να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είχαμε και επιτυχίες, πρέπει να το πω. Να αναφέρω καταρχάς την κοινωνική διάσταση της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ένα παιδί που δεν ήταν πολύ αγαπημένο επί πολλές δεκαετίες που πέρασαν. Υιοθετήσαμε το, η βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε μια πρώτη εμφάνισή μου σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν Υπουργό Εργασία επί Λουξεμβουργιανής ε, Προεδρίας, την ομιλία που κάναμε. Πριν εγκριθεί ε, η βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων, είχαμε δρομολογήσει την οδηγία για τις αποσπάσεις. Και αντίθετα από τις προσδοκίες, καταφέραμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τα οδηγήσουμε να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταρχήν θέσπισε την αρχή ότι για την ίδια ε, θέση εργασίας και το ίδιο έργο και την ίδια θέση πρέπει να υπάρχει ίδια αμοιβή. Εάν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη που θα ευημερήσει πρέπει να ακούσουμε αυτούς που εργάζονται. Αλλιώς θα κάνουμε σφάλμα θα πρέπει να είναι η Ευρώπη μια Ευρώπη που είναι η Ευρώπη και για τους εργαζομένους. Άλλη επιτυχία πιστεύω. Η Ελλάδα. Μιλάω γι' αυτό διότι με απασχόλησε πάρα πολύ και με ανησύχησε πάρα πολύ το θέμα. Ξαναδώσαμε στην Ελλάδα την αξιοπρέπεια που της αρμόζει. Πολύ συχνά και επί πολύ μεγάλο ε, μακρό διάστημα ποδοπατήσαμε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και θέλουμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στην τάξη τους. Να ξαναδώσουμε σε αυτό το λαό όλους τους τίτλους αξιοπρεπίας και ευγενία που του αξίζει. Λοιπόν, ε, θέλαμε να κινηθούμε υπέρ της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάμαι μακρές ε, νύχτες με τις κυβερνήσεις Σαμαρά, Τσίπρα και τώρα του ε, κυρίου Μητσοτάκη όταν δεν είχε αναλάβει ακόμα προσπαθήσαμε να επιλύσουμε τα ελληνικά προβλήματα, το ελληνικό πρόβλημα και πολλοί, πολλές ήταν οι κυβερνήσεις που δεν ήθελαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα της Ελλάδας. Θυμάμαι τα τηλεφωνήματα πάντα πολλών πρωθυπουργών που μου έλεγαν ασχοληθείς εσύ με τα θέματά σου. Είναι θέμα των χωρών να ασχοληθούν με το ελληνικό πρόβλημα. Ενώ εγώ είχα την αφελή αντίληψη ότι θα έπρεπε να σεβαστούμε τις συνθήκες. Και τι ήταν οι συνθήκες. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον ε, της Ευρώπης να αποφευθεί από σύνθεση της Ευρωζώνης. Λοιπόν, Σωστά κάναμε αυτό που κάναμε. Είχαμε δίκιο. Η Αφρική. Η Αφρική Σαν Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τους γείτονές μας, πρώτους γείτονές μας που είναι οι Αφρικανοί. Είναι μια ήπειρος που χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. αλλά όχι μόνο ε, την ε, φιλανθρωπία μας. Φιλανθρωπία είναι παλιά αντίδραση των Ευρωπαίων, ενώ σήμερα Πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε μια συνεργασία ισότιμη μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, επενδύοντας στην Αφρική, δημιουργώντας θέσεις εργασία στην ε, Αφρική. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητο των δράσεών μας, να μην βλέπουμε την Αφρική μόνο μέσα από το πρίσμα της κρίσης της προσφυγικής. Πληγώνουμε την περηφάνεια των Αφρικανών όταν βλέπουμε τη σχέση με την Αφρική μόνο από το πρίσμα αυτό ε, των προσφύγων. Θα πρέπει να κάνουμε επιτόπου αυτό που ε, πρέπει για να μην αναγκάζονται οι ατυχείς να περνούν του ωκεανούς. Ε, τώρα για τους, ε, είχαμε επιτυχίες όσον αφορά τους πρόσφυγες. Είναι καλύτερος ο απολογισμός από ό,τι μπορούσαμε να πιστέψουμε, αλλά μπορούσαν καλύτερα τα πράγματα. Το Συμβούλιο, όπως έκανε το Κοινοβούλιο, είχε συμπορευτεί με τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους νομοθέτες. Πρώτα απ' όλα για τη μετεγκατάσταση τον Μάρτιο του 2015 είχαμε κάνει πρόταση και μια άλλη τον Απρίλιο του 2016 όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Μιλείς όμω όμως ότι χάρη στην Ευρώπη καταφέραμε να σώσουμε στη Μεσόγειο 760.000 χιλιάδες ε, ανθρώπους που αυτοί είναι λιγότεροι νεκροί ε, χάρη στη δράση που έκανε η Ευρώπη. 76.000 μάλλον. Οι μόνοι επιβιώσαντες, οι μόνοι αυτοί που χειροκροτούν. Είχα πει ε, το Μάρτιο του 2015 αυτά που κάναμε όσον αφορά τους πρόσφυγες. Και όρθιοι με χειροκρότησαν στο κοινοβούλιο. Και, και γιατί με χειροκροτείτε, είπα. Είσαστε σίγουροι σε δύο χρόνια ότι πάντα θα με χειροκροτείτε. Τα χειροκροτήματα ήταν πιο ισχνά τα επόμενα χρόνια, διότι σε πολλές χώρες η εσωτερική πολιτική επεκράτησε επί της βασικής αλληλεγγύης που θα έπρεπε να εφαρμόζαμε. Ασχολήθηκα πολύ, περισσότερο από ό,τι νόμιζα όταν έφτασα να είμαι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ασχολήθηκα περισσότερο με το διεθνές εμπορίο, ένα δύσκολο θέμα, ε, άκρος επίμαχο σε όλες τις χώρες μας και πολύ συχνά υπήρχαν πολλά επιχειρήματα σωστά κατά των εμπορικών συμφωνιών που συνήπτονται βιαστικά. Το αλλάξαμε αυτό, συνήψαμε 15 συμφωνίες εμπορικές διεθνείς. Σήμερα έχουμε εμπορικές συμφωνίες με 60 χώρες. Αυτό αντικατοπτρίζει 40% του πλούτου του παγκοσμίου και αυτές οι συμφωνίες μας βοηθούν να είμαστε παρόντες στο διεθνές προσκήνιο ε, μια στιγμή όπου οι ΙΠΑ γυρνούν την πλάτη τους στην πολυμερή προσέγγιση, άρα και στην οργανωμένη αλληλεγγύη με τους άλλους. Η μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρώπης παραμένει το γεγονός ότι μπορέσαμε να διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται 60 πόλεμοι παγκοσμίω. Καμία πολεμική σύγκρουση όμως δεν λαμβάνει χώρα στο έδαφος της Ένωσης που υπήρξε θέατρο ε, των πιο αιματηρών πολέμων και τον προηγούμενο ε, αιώνα μάλιστα. Ε, καταφέραμε να διατηρήσουμε την ειρήνη και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γνωρίζω ότι οι νέοι δεν ενθουσιάζονται σκεπτόμενοι τη διατήρηση της ειρήνης. Σκεφτόμαστε εμείς. Πρέπει όμως να μιλήσουμε με τους νέους Γι' αυτό το μεγάλο δίλημα της Υπήρου μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Πρέπει να πλησιάσουμε τους πολίτες και να δούμε πώς, εκλαμβάνουν, ε, πώς προσλαμβάνουν την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και διεθνές επίσης. Πρέπει να τους ε, μιλάμε για τον πόλεμο και την ειρήνη στους ε, νέους. Σε 20 χρόνια ε, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται τον πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τη μνήμη, γιατί αλλιώς θα ξεχάσουμε τι σημαίνει πόλεμος. Γι' αυτό συζητώ πάντα για πόλεμο και ειρήνη με τους νέους. Αλλά δεν φτάνει να εξηγούμε πρέπει στους ε, νέους να εξηγήσουμε και τις προοπτικές της Ευρώπης, το μέλλον της Ευρώπης. Είμαστε η μικρότερη Ήπειρος. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Είμαστε πολύ μικροί ως Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Στην πολιτική συνδυάζομαι την ε, γεωγραφία και τη δημογραφία. Δεν μπορεί να διαχωριστούν αυτά τα δύο. Ε, δεν θα εξαλειφθούμε, αλλά ε, ο αριθμός μας μειώνεται. Στο τέλος αυτού του αιώνα, 4% 10, επί των 10 δις θα είναι Ευρωπαίοι πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας τον κίνδυνο που υπάρχει ότι μπορεί να χάσουμε ε, ένα κομμάτι από την δύναμή μας. Οι εξελίξεις αυτές είναι ε, μη αναστρέψιμες και θα πρέπει να ε, δούμε την Ευρώπη εν συνόλο και όχι μέσα από το εθνικό πρίσμα και μόνο. Θα ήταν λάθος αυτό. Και σε σχέση με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε ε, νυφάλιες και σωστές αποφάσεις το ζήτημα της ειδική πλειοψηφίας ε, στις αποφάσεις του Συμβουλίου επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής είναι σημαντικό. Όχι, επειδή, όχι επί όλων των θεμάτων, αλλά θα πρέπει να παίρνει θέση περισσότερο η Ευρώπη. Στην, ε, ε, επισκέφθηκα τον πρόεδρο Τραμπ για να συνομιλήσω μαζί του σχετικά με την αποτροπή του εμπορικού πολέμου. Τα κατάφερα. Πώς. Ο Τραμπ έκανε μια μεγάλη εισαγωγή, το συνηθίζει αυτό, και εκεί παρευρίσκονταν ε, στη συνάντηση και διάφοροι σύμβουλοι ε, εγώ του είπα θα πρέπει να, αυτά που μας λέτε να τα εξηγήσω ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στους ε, ε κρατών και κυβερνήσεων διότι η Κομισιόν δεν μπορεί παρά δεν, δεν δρά διαφορετικά. Και τότε φάνηκε ότι η απάντησή μου του έκανε εντύπωση. συμπερασματικά. Δεν αποχωρώ θλιμμένος, ούτε βέβαια υπερβολικά ευτυχής, αλλά έχοντας τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι ε, προσπάθησα πολύ. Όπως και οι συναδελφοί μου. Τα τελευταία πέντε χρόνια ε, περηφανεύομαι να πω ότι Αποτέλεσε ένα μικρό κομμάτι ενός μεγάλου συνόλου που είναι η Ευρώπη. Και έδωσα μάχη με όλες μου τις δυνάμεις ε, τον εθνικισμό. Ζήτω η Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ. Και τώρα θα ακούσουμε κάποιες παρατηρήσεις από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων. Κύριε Βέμπερ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε lieber Αγαπητέ Πρόεδρε Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, η πολιτική ζει μέσα από την αλλαγή. Σήμερα ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ένας μεγάλος Ευρωπαίος, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, εγκαταλείπει ε, το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Οι χριστιανοδημοκράτες σε ευχαριστούν θερμά για την προσφορά σου όχι μόνο τα προηγούμενα πέντε χρόνια, επί ε, πριν από 36 χρόνια συζήτησες για την ε, ε, νομισματική ένωση, διαπραγματεύτηκες με την Ιρλανδία, ε, πολλές φορές ε, έκανες διαπραγματεύσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας ως Λουξεμβούργιος και Πάντοτε σε απασχόλησε η δημοκρατική πορεία της Ευρώπης. Μαζί με τον Μάρτιν Σούλτς παραμένετε ιδρυτές αυτής της δημοκρατικής Ευρώπης. Ε, κυρίως ε, γνωρίζεις να, να κάνεις σωστούς συμβιβασμούς. Πολλές φορές διαμεσολάβησες για να συμφιλειωθούν ε, με, ε, διαφορετικά μέρη μεταξύ τους. την ε, Επιτροπή σου την ε, ανέφερε σε Επιτροπή της τελευταίας λύσης. Ε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα κατά την προηγούμενη πενταετία. Εμεί δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι λύσαμε τα προβλήματα, αλλά εμψυχωμένοι συνεχίζομαι αντιμετωπίστηκαν προβλήματα μέσα σε μια πενταετία που θα έπρεπε να απασχολήσουν ε, την Επιτροπή για μια είκοσα αιτία. Οι ευκαιρίες ε, αξιοποιήθηκαν. Σήμερα η Ευρώπη είναι σε καλύτερη ε, θέση από ό,τι παλιά. Υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκαν εμπορικές συμφωνίες, τίναμε χείρα βοηθεία στην Αφρική αντιμετωπίζω με τον Brexit είναι μια περισσότερο ευημερούσα Ευρώπη, πιο σίγουρη Ευρώπη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα σημαντικά θέματα. Νομοθετήματα είναι το ένα. Η πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων είναι κάτι διαφορετικό. Αν δούμε την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, ανέφερε σε την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες χώρες, τα τελευταία χρόνια με τη δική σου εφαρμογή των κειμένων μάθαμε ότι πίσω από κάθε νομοθέτημα κρύβονται άνθρωποι και πρέπει να τους σεβαστούμε και να τους ε, πάρουμε στα σοβαρά. Αυτό το κατάφερες ε, εσύ περισσότερο από κάθε άλλον. Ένα άλλο που συγκρατώ είναι ότι η Ευρώπη από πολλούς αντιμετωπίζεται ως Ευρώπη των αγορών, ε, του χρήματος. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των αγορών, αλλά υπέρ της κοινωνικής ε, οικονομίας. Ε, είσαι παιδί ενός ε, ανθρακορίχου και εγνώριζες πολλά θέματα πρακτικά όταν πήγαινες για τις συνομιλίες στον Ταβός έβαλες πάρα πολλά θέματα σημαντικά ε, για τους ε, ανθρώπους ε, στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, δεν συμβιβάστηκες ποτέ εις ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αξίες. Η Ευρώπη το, της ισότητας, της προστασίας των μειονοτήτων, η Ευρώπη της ελευθερίας. Γι' αυτή την Ευρώπη έδωσες μάχες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, χωρίς συμβιβασμούς. Σε ευχαριστούμε για, αυτό. Η ευρωπαϊκή ιδέα απέκτησε νέο νόημα. Οι λαϊκιστές της αριστεράς και της δεξιάς αντιμετωπίστηκαν αποφασιστικά από εσένα. Ε, ο αυξημένος, ε, το αυξημένο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για την Ευρώπη είναι εν μέρη και δικό σου έργο. Ε, εμείς ως ΕΛΚ θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Τέλος, Ζαν Κλόντ, η ομάδα σου, η ομάδα του ΕΛΚ είναι περήφανη για τη θητεία σου. Ε, μας προφύλαξες από πολλές ζημιές ε, στην Ήπειρό μας. Ε, είναι, ε, είμαστε περήφανοι που σε έχουμε στις γραμμές μας συνάδελφοί σου ε, γνωρίζουν ότι με τον ε, Ρομπέρτ Σουμάν, τον Αλτζίντε ε, Τεγκάσπερη και τους άλλους πατέρες της Ευρώπης και εσύ συνέβαλες στην ευημερία της Ευρώπης. Αυτή είναι μια σχέση αγάπης, είπες εσύ. δεν είναι μόνο μια σχέση αγάπης που μπορεί να κρατήσει λίγο, είναι ένας δεσμός που κρατάει μια ολόκληρη ζωή και θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε επιτυχίες ε, με βάση τις ιδέες για τις οποίες ε, ε, επάλεψες. Σε ευχαριστούμε ολόκληρη η ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Βέμπερ. Πρόεδρε Γκαρθία Πέρες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, για να ξέρουμε μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πώς φτάσαμε εδώ. Δεν ήταν εύκολη πορεία και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Γιούνκερ. Πριν από πέντε χρόνια εσείς ε, μας προτείνατε ένα νέο θεματολόγιο. Λεγόταν μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Αλλά αυτή η νέα αρχή έμεινε στα μισά του δρόμου συνειδητοποιούμε ότι εσείς ε, κάνατε προσπάθειες. Εσείς προσπαθήσατε να αποστασιοποιηθείτε από τις πολιτικές λιτότητας ε, και τις αυστηρές πολιτικές που μας είχε επιβάλει ο πρόεδρος Μπαρόσο. Και πάντα είχατε τη στήριξη της πολιτικής μας οικογένειας ε, στη στάση σας αυτή. Οι συνέπειες της κρίσης μας έπληξαν όλους και σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν μπορέσαμε να λάβουμε τις ριζοσπαστικές αποφάσεις που χρειαζόντουσαν ώστε να αλλάξουμε πορεία. Ελπίζω στη νέα θητεία να μπορέσουμε να το κάνουμε. Όταν εσείς φτάσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνατε ένα σύνολο θεμάτων και καταφέρατε να ε, προτείνετε το 90% εξ αυτών, αλλά εγκρίθηκαν μόνο οι μισές. Και περισσότερες έμειναν στο σιρτάρι και κάποιες από αυτές ήταν πολύ σημαντικές. Ορισμένες φορές η αποτυχία δεν οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην έλλειψη ε, για συνεργασία των κρατών μελών της Ένωσης. Μας προτείνεται ένα θεματολόγιο για απασχόληση, ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και είναι αλήθεια ότι ήταν φιλόδοξο και δύσκολο το έργο σας, αλλά οι συνέπειε ε, τη πιο αυστηρή ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που βίωσε ποτέ η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι. Και υπήρχε διαχείριση με πολύ μεγάλη έλλειψη αλληλεγγύη και τη δυσάρεστη έκπληξη του Brexit. Δεν είναι λίγο αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε τι κάναμε λάθο για να μην ε, διαπράξουμε τα ίδια σφάλματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πάντα με είχατε στο, στο πλευρό σα για τι αξίε και τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σοσιαλδημοκράτε δράσαμε με ευθύνη και υπερασπιστήκαμε ανα πάσα στιγμή το ευρωπαϊκό σχέδιο, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ε, ε, ακάματη εργασία του Φραν Τίμερμαν ε, για τι κοινέ αξίε και αρχέ, τη μάχη κατά του εξτρεμισμού, και των ακραίων θέσεων και σίγουρα αυτό ενίσχυσε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να πετούμε την ίδια δέσμευση για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα είχατε επίση στο πλευρό σα αναζητώντα μια λύση για την μεγάλη μεταναστευτική κρίση. Σα ευχαριστούμε για την προσπάθειά σα ε, για να μπορέσουμε να βρούμε μια απάντηση η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ευθύνη των κρατών μελών. Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να ε, τα δεχτεί αυτά το Συμβούλιο, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να καταφέρουμε να ε, ανανεώσουμε ανανεώσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ήμασταν στο πλευρό σα ε, για να ε, ανταποκριθούμε στις επιθέσεις ε, στην πολυμορφία. Θέλουμε να έχουμε ένα πιο δίκαιο εμπόριο και η Ευρώπη να μιλάει με μία μονοφωνή και εσείς ε, δώσατε μάχη και είχατε μία συμμαχία με την ύπατη εκπρόσωπο ε, την κυρία Μογκερίνη και έτσι θεμελιώσατε όχι μόνο μια νέα συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά εμβαθύναμε και σε μια ιστορική συμφωνία με το Ιράν. Αυτό που δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε παρκώς είναι τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και την οικονομική μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ζητήσαμε πριν από πέντε χρόνια, εσείς καλωσορίσατε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο των Επενδύσεων, που ήταν ο σπόρος για το European Green Deal και το σχέδιο επενδύσεων που θέλει να προωθήσει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό δεσμευόμαστε με περισσότερη ενέργεια, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Το σχέδιο Μοσχοβησί ήταν θεμελιώδε, ώστε να έχουμε ευελιξία στο Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Ε, σε απάντηση στην παράλογη λιτότητα και στην αυστηρότητα που επέβαλε η δεξιά. Κύριε Μοσκοβισή, σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Είναι απαράδεκτο το Συμβούλιο να έχει απορρίψει τόσες προτάσεις ε, για να βελτιώσουμε τη φορολογική δικαιοσύνη, ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και όχι μόνο ε, να πληρώνουν οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή σας, κύριε Γιούνκερ, ανταποκρίθηκε και στα αιτήματά μας για έναν κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά αυτό είναι μόνο η εκκίνηση. Θέλουμε ο πυλώνας αυτός να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα, να υπάρχει καθολική πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και να υπάρχει συλλογική προστασία, να ε, εκριζώσουμε την παιδική φτώχεια και να υπάρχει συμφωνία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Σε θέματα ισότητας υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, πράγματι και σήμερα μετά από την πρόταση και την ανακοίνωση της Επιτροπής σας για το στόχο που επέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσουμε στο 40% των γυναικών σε θέσεων ε, διευθυντών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι αυτή είναι εξαιρετική είδηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορούσε να μας αποχαιρετήσει με καλύτερο τρόπο, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη που είναι χωρίς ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την πολιτική μας ομάδα, αλλά και για μένα προσωπικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που κάνατε επί του θέματος. Δυστυχώς, οι συντηρητικέ δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν επέτρεψαν μεγαλύτερη πρόοδο. Δεν φταίτε εσεί, κύριε Γιούνκερ, δεν σα κατηγορούμε εσά. Σα ευχαριστούμε για τον ευρωπαϊκό ενθουσιασμό σα και το χιούμορ σα. Και με μία φράση θα τελειώσω με αυτό που είπατε εσείς. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει μάχη κατά του εθνικισμού γιατί η Ευρώπη είναι ένα σχέδιο συμβίωσης, είναι ένα σχέδιο ειρήνης και σήμερα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τη δέσμευσή σα. Έχετε τον πλήρη σεβασμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιούνκερ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε Τσόλο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγαπητέ Ζαν Κλοντ, δράτω με αυτές τις σημαντικές στιγμής για να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για τις δράσεις σας ως επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά για την καριέρα σας πεπισμένου Ευρωπαίου. Δώσατε πολλά μαθήματα σχετικά με το τι σημαίνει ένας πραγματικός Ευρωπαίος. Σας ευχαριστώ για αυτό. Στη θητεία σας έπρεπε να είστε τη σελίδα της οικονομικής κρίσης, να αντιμετωπίσετε το Brexit και την κρίση τη μεταναστευτική μπορέσατε να διατηρήσετε την Ευρωπαϊκή Ενότητα και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος ομόφωνα εδώ σας ευχαριστεί διότι αυτή η ενότητα είναι το πιο πολύτιμο κοινό αγαθό. Κάποιοι αποκάλυψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη τελευταία ευκαιρία. Τώρα, μια άλλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθέστη τη και οι αντιευρωπαίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν και ήλπιζαν. Θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη που είναι χρήσιμη για του πολίτε μα. Αυτό είναι στο επίκεντρο προσπαθειών Ευρωπαϊκής, ε, του Κοινοβουλίου και θα έχουμε μια ευκαιρία μέσω τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, λοιπόν, πολλά επετέφθησαν κατά τη διάρκεια αυτών των ε, ετών τη θητεία σα όταν ήσασταν επικέφαλή Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Μπορώ να παραθέσω πολλά παραδείγματα συγκεκριμένα, αλλά θα σταθώ πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο Juncker. Δεν μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό. Είχε κατακριθεί στην αρχή, είχε επικριθεί, παρόλα αυτά επέτρεψε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτά. Ε, στήριξε πολλές μικρές, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έδειξε το πρόσωπο της αποτελεσματικής Ευρώπης που μπορεί να ε, δρομολογήσει καινοτόμα προγράμματα. Ήταν πιο πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπατε στην παρέμβασή σας, και να ανοίξατε το δρόμο, πιστεύω, που θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε να γίνει πιο πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πολιτικής στα ευρωπαϊκές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο μέσω ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μεταξύ των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων για να οικοδομήσουμε σταδιακά αυτή την Ευρώπη που είναι στην καρδιά των προσπαθειών σας. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Jean-Claude Juncker. Ευχαριστούμε όλη την Ευρωπαϊκή σας Επιτροπή διότι δείξατε, αποδείξατε ε, τι είναι δουλειά για την Ευρώπη, τι είναι να καταβάλλετε προσπάθειε για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Λάμπερτς, έχετε εσείς το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ζων Κλόντ, εν ονόμα της ομάδας των Πρασίνων, θέλω εδώ ε, να σας ευχαριστήσω για τη Μετά πέντε χρόνια, πέντε χρόνια που πέρασαν, ε, ψήφισα για σας τότε εδώ και πέντε χρόνια να είσαστε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έκανα όταν είσαστε εκείνος όταν το μεγάλο δουκάτο ότι την διακυβέρνησή σας έγινε ε, κάπως ε, φορολογικός παράδεισος στο Λουξεμβούργο. Ε, ίσως τελικά ε, επειδή ξέρατε από αυτά γίνατε ο καλύτερος ε, προστάτης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λοιπόν, πρέπει να γνωρίσουμε ότι στη θητεία σας λοιπόν η φορολογική δικαιοσύνη προωθήθηκε αλλά παρέμεινε να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο εμπόδιο το πείσμα των κρατών μελών που ειρνούνται κάθε εναρμόνιση φορολογική. Αυτό το εμπόδιο μπορέσατε να το επερκεράσετε μέσω του άρθρου 116 τη συνθήκη. αλλά δεν είχα την τόλμη να το κάνετε τελικά. Για να είμαι ειλικρινή, θέλατε κοινωνική δικαιοσύνη και τελικά είχατε το πρόσωπο ε, χριστιανοδημοκράτη που τελικά είχατε μπει στα πλαίσια του ΕΛΚ. Είχαμε την οδηγία στου προσωπικού εργαζομένου, θέλαμε μια ευρωπαϊκή αρχή που προτείνατε για την εργασία που ήταν και ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά διεμφισβήτητα ήταν επιτυχίες που μπορούν να μπουν στον απολογισμό σας και των συναδέλφων σας. Ειδητήσετε μία λιγότερο άκαμπτη ιδεολογική προσέγγιση των ευρωπαϊκών κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης ε, μειώνοντας κάπως ε, τη λιτότητα που θα ήταν τυφλή και κοφή ε, στις απαιτήσει της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Λόγω ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφίστη προσπαθειών ούτω ώστε οι Ευρωπαίοι να βρουν συλλογική και αλληλέγγυα απάντηση στο, προς, στο πρόβλημα του ασύλου και τη μετανάστευση. Αλλά και σε αυτό το σχέδιο ε, πρόβαλε αντιστάσει στο Συμβούλιο και λυπούμε που ο κ. Στούσκ δεν είναι εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, και έδειξε μεγάλο πείσμα και τελικά διατήρησε αυτή την Ευρώπη φρούριο. Αν αυτή η κοινωνική σα είναι ένα η υπερβαντική σα συνείδηση ε, πρέπει να προωθηθεί. Ο κοινό μα οίκο καίγεται από ένα κλίμα που αλλάζει, βιοπικιλότητα που καταραίει και από πόρου που εξαντλούνται. Στο επίκεντρο αυτή τη πυρκαγιά, μια παγκοσμιοποίηση όπου οι συνθήκε ε, των ελευθερών συναλλαγών την του. και ε, οι επενδυτέ διακινούν τα κεφάλαιά του και οι φορολογικές δημοκρατικές προδιαγραφές τελικά δεν εφαρμόζονται σωστά, ε, δεν είναι αρκετά περιοριστικά αυτά τα μέτρα Λοιπόν, ε, καμία δεκαπενταριά ε, συμφωνίε έχουν συναυθεί με διάφορε χώρε. Υπερασπιστήκατε εκείνη αγροτική πολιτική που παράγει περισσότερο παρά τι φιλοδοξίε για την βιοπικιλότητα και την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Παρά τι υποσχέσει σα και λυπούμεθα γι' αυτό ει βάθο, διότι κάνατε υποσχέσει στην ομάδα μα εδώ και πέντε χρόνια, μπλοκάρατε κάθε πρόοδο όσον αφορά την απαγόρευση των ενδοκρινικών διαταρακτών και δεν εκδημοκρατήσατε την ε, έγκριση των ε, διαφόρων ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Υποστηρίξατε το big business. Ε, προστατεύσατε ε, το επαγγελματικό απόρριτο ένθερμα και δεν προστατεύσατε τις πληροφοριοδότες κοινού συμφέροντος. Επαρκώς. Λοιπόν, έχουμε ανάμεικτες αναμνήσεις πενταετίας σας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταβατική που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει πλήρως τα υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μα λέγατε ότι ήταν τελευταία ευκαιρία, ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Τελευταίας Ευκαιρίας. Ε, τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου σας διέψευσαν ευτυχώς. Οι πράσινοι ε, ε, έπαιξαν το ρόλο τους στην αλλαγή που έρχεται. Η λογική της εθνικής προτίμησης τελικά δεν ε, νίκησε και όπως και εσείς θα την καταπολεμήσουμε αυτή την προσέγγιση εθνικιστική. Όμως δεν απομακρυνθεί ο κίνδυνο εκείνοι που θα σας ακολουθήσουν πρέπει να το κάνουν αυτό. Και η Πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δεχθεί τη δική σας, όλοι αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία εάν όπως το θέλετε και εσείς και εμεί θέλουμε να συμφιλιώσουμε όλου του Ευρωπαίου, άντρε και γυναίκε με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπενθυμίζω πρώτη εμπειρία, πρώτο πείραμα στον κόσμο για μια δημοκρατία υπερεθνική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τζάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε Γινκέρ, πριν από πέντε χρόνια όταν εσείς ε, ήσασταν ε, εδώ στην ε, Ολομέλεια. Εγώ είχα εκφράξει μεγάλες αμφιβολίες για το κατά πόσον εσείς θα μπορούσατε να είσαστε ο σωστός άνθρωπος για αυτή την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Σας αφήσαμε όμως ε, το δικαίωμα να έχουμε και κάποιες αμφιβολίες. Πρέπει να πω μετά χρόνια μετά ότι η αμφιβολία επιβεβαιώθηκε. Εσείς μας παραδίδετε μια Ευρώπη η οποία είναι χειρότερη από αυτή που αναλάβατε πριν από πέντε χρόνια. Μια Ευρώπη διαιρεμένη, μια Ευρώπη αδύναμη, μια Ευρώπη άρρωστη η οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και στα τρία ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και σας ζητήσαμε να επιλύσετε το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης και το πρόβλημα της ασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας. Η Επιτροπή σας και η θητεία της αυτή την πενταετία απέτυχε και στους τρεις αυτούς στόχους. Και φυσικά δεν πρέπει να αναζητούμε τα αίτια εκτός των θεσμικών οργάνων. Τα αίτια είναι εσωτερικά. Τα αίτια είναι οι λανθασμένες πολιτικές τις οποίες προωθήσατε, επαναλαμβάνοντας λάθη τα οποία είχαν διαπραχθεί και από την προηγούμενη Επιτροπή. Εσείς αναφερθήκατε για τις υποτιθέμενες επιτυχίες της Επιτροπής σας, αναφερθήκατε στην ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη είναι ασφικτική και η Ευρώπη χάνει έδαφος σε σχέση με τις υπόλοιπες ε, χώρες εκτός των ε, συνόρων μας. Δεν αναφερθήκατε στη ε, στον εκβιομηχανισμό και κάποιες επιχειρήσεις έχουν αποτύχει και δεν λειτουργούν πλέον. Αναφερθήκατε σε επενδύσεις και παραδεχτήκατε ότι είχατε 140 επιπλέον εκατομμύρια, δισεκατομμύρια επενδύσεις. Ε, αλλά μας είχατε υποσχεθεί 315 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το 50% αυτού που υποσχεθείτε μπορεί να θεωρείται επιτυχία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πελίτε οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι που εσεί θα μπορέσετε να απολαύσετε επιπλέον τη σύνταξή σα, διότι η Επιτροπή σα ήταν η χειρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων ετών στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχετε και μια παρηγοριά, διότι εγώ πιστεύω ότι ο διάδοχό σα θα μπορέσει σίγουρα να τα κάνει χειρότερα. Δεν είναι βέβαια καλό το νέο αυτό για του Ευρωπαίου πολίτε και εμεί φυσικά δεσμευόμαστε ώστε τα τεράστια ολέθρια σφάλματα τα οποία διαπράξατε τα τελευταία χρόνια να μην ξανασυμβούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο κύριος Λεγκούτκο. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσω την αφοσίωσή σας στο δημόσιο ε, αξίωμά σας πρέπει να επενεθείτε γι' αυτό, όπως πρέπει να εκτιμηθεί και το έργο των συνεργατών σας για την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς, την ε, ισχυροποίηση των ενεργειακών, ε, του ενεργειακού εφοδιασμού και ε, τα καλά σχέδια για την ενίσχυση των μικρομεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων σε αρκετά σημεία Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Όμως η θητεία σας χαρακτηρίστηκε και από αρκετές απογοητεύσεις. Ε, η απώλεια ενός μεγάλου κράτους μέλους που ασκεί τεράστια επιρροή σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια ιστορική απογοήτευση και μη μας πείτε ότι δεν φέρετε την ευθύνη γι' αυτό. Θα έπρεπε να την φέρετε. Αυτό που επίσης με ανησυχεί είναι ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ε, ε, ε, υπήρξε έναυσμα για προβληματισμό όπως θα έπρεπε για να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια. Ο κύριος ε, Μπαρνιέ μίλησε για προβληματισμό ε, σήμερα το πρωί, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν και όχι μετά το Brexit. Ανταυτού είχαμε μια πολιτική που βάθινε της διαιρέσεις και επιδίνωσε τα προβλήματα. Η απερχόμενη επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε, επιδίωξε ε, ε, στηρίχθηκε στις περισσότερα δημοκρατικά ε, εκλεγμένες κυβερνήσεις και εσείς ε, επιτείνεται τον διχασμό μεταξύ κρατών μελών ε, τονίζοντας ε, παραβιάσεις και αγνοώντας άλλες. Υπήρχαν χώρες που παραβίαζαν τους κανόνες για τη μετανάστευση και μετά ακολουθήθηκε μια διαιρετική πολιτική στα κράτη-μέλη επιβάλλοντας επιχειρώντας να επιβάλλουν κανόνες που τα κράτη δεν ήθελαν. Είναι ε, σημαντικό η Επιτροπή να συνενώνει και όχι να διαιρεί τα κράτη-μέλη. Και η απερχόμενη Επιτροπή, λυπούμε που το λέω κυρία Γιούγκερ, είναι η πρώτη που έκανε τα περισσότερα για να ε, απομακρύνει τα κράτη το ένα από το άλλο παρά να τα συνενώσει. Πρόεδρε Ομπρή, έχετε το λόγο. Κύριε Πώ να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον απολογισμό χωρί να παραθέσουμε τον ατέρμονα κατάλογο σκανδάλων των φορολογικών παραδείσων που στόλισαν ε, τι εξελίξει ε, Panama Papers και λοιπά και τα Lux Leaks, ε, των οποίων ε, είσαστε εμπλεγμένος εσεί στη χώρα στο Λουξεμβούργο που τελικά είναι παράδεισος φορολογικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής ε, έπρεπε να επιτευχθεί και πάση προσπάθειε κάποιων επιτρόπων που χαιρετίζουμε τη θητεία τους είναι σαν ζητούσαμε από τη Μονσάντο να θέσει τέρμα στα παρασιτοκτόνα. Ήταν στο αρχηγό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο κοινωνικό πυλώνα, άρα παραμένει αποτυχία. Πού είναι ο ελάχιστος ευρωπαϊκός μισθός που μας υποσχεθήκατε. Ο απολογισμό, κύριε Γιούνκερ, όσον αφορά το κλίμα, είναι απογοήτευση. Δεν αναλάβατε υποχρεώσει από αυτού εδώ και πέντε χρόνια. Έτσι δεν είναι. Και με οι συνθήκες ελεύθερων συναλλαγών τελικά δεν το έλαβαν αυτό υπόψη. Αυτός ο απολογισμό για τις διασωμένες, τις ε, που σώθηκαν. Έχουμε 16.000 νεκρούς όμως, που θα πρέπει να είναι ντροπή, όνειδος για μια Ευρώπη που μεταμορφώθηκε σε κάστρο. Ο απολογισμό σα είναι ένα κλείδωμα δημοκρατικό τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει δικαίωμα πρωτοβουλία για το Κοινοβουλίο και ελπίζω ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα το προωθήσει. Οι αντίπαλοι σα όπω είπατε τελικά, είπαν ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική επιλογή κατά των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και εμεί πιστεύουμε το αντίθετο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκέ συνθήκε χωρί δημοκρατική επιλογή. Κατά, στο τέλο τη θητεία σα, κύριε Γιούνκερ, επιτέλου εξυπηρετήσατε τελικά τι αγορέ στη θητεία σα και απογοητεύσατε του Ευρωπαίου συμπολίτε. Εμεί είμαστε υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σα ευχόμεθα έξοχη σύνταξη. Και γι' αυτό, όπω και έχουμε για εσά ένα δωράκι για να επιστρέψετε στο φορολογικό σας παράδεισο. Οι φίλοι σας, οι πολυεθνικές που βοηθήσατε στα LuxLeaks σας εύχονται ε, μια ευτυχή ε, σύνταξη με αυτό το δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Γιούνκερ η θητεία σας και αυτή της Επιτροπής σας ολοκληρώνεται. Είναι ο χρόνος λοιπόν να κάνουμε απολογισμό. Ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου δυστυχώς ε, δεν μπορώ να σας βαθμολογήσω για κάθε μάθημα γιατί θα ήσασταν ε, ε μεταξυταστέως τα περισσότερα. Το σχέδιο επενδύσεων λοιπόν με το όνομά σα, το σχέδιο Juncker, είναι ένα σχέδιο το οποίο αντί να ε, στοχεύσει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στην ενεργειακή αποδοτικότητα, επενδύει σε ορυκτά καύσιμα ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι στην ενέργεια. Από τα 195 έργα τα οποία εγκρίθηκαν το 2015, τα περισσότερα αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό άργορο. Το ίδιο και για το 2019. Έχουμε 55 τα οποία είναι για ορυκτά καύσιμα. Έτσι θέλουμε πραγματικά λοιπόν να κάνουμε την ενεργειακή μετάβαση σε μια ιστορική εποχή για την ε, κλιματική αλλαγή. Εσείς έχετε καθυστερήσει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της και φυσικά αυτό θα πρέπει να το εξηγήσετε και στους νέους που διαδηλώνουν στους δρόμους ε, σε όλη την Ευρώπη και στις επόμενες γενναίες. Αυτές τις μέρες συζητάμε, όπως γνωρίζετε, ένα νέο ε, σχέδιο επενδύσεων, αυτή τη στιγμή ε, βιώσιμων επενδύσεων, ελπίζουμε, το οποίο πρότεινε η Πρόεδρο Βαντερ Λάιεν. Ε, πολλά ευρώ, δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική ευρώ ε, αλλαγή, συγγνώμη. Ελπίζω όμως ε, να μην ε, ε, έχουμε τα λεγόμενα σχέδια τα οποία προωθήσατε κι εσείς με το σχέδιο Γιούντερ και για τα οποία το ελεγκτικό συνέδριο έχει ήδη εκφράσει αμφιβολίες μου. Και θα ήθελα κι εσείς να ζητήσετε συγκεκριμένε εγγύησεις από την πρόεδρο Βαντερ Λάιον ώστε αυτό το νέο Green Deal να προσφέρει πόρους για να σιώσουμε τον πλανήτη. Χρειαζόμαστε πράσινες επενδύσεις και όχι λογιστικά αλλά Juncker. Στο τέλος της συζητήσεως, το λόγο έχει ο κύριο Γιούνκερ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν στη συζήτηση, κυρίως εκείνους που τοποθετήθηκαν επενετικά και ο κύριος Τζάνιος μελετήσει καλύτερα το χαρτοφυλάκιό του Αλλιώς δεν θα απαρέθετε τόσο ψευδή νούμερα, αναλυθή νούμερα. Πρόεδρε Γιούνκερ, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την παρουσία σας, για τις προσπάθειές σας, για την πράσπιση του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους και εν ονόματι του Κοινοβουλίου σας Απευθύνω την ευγνωμοσύνη μας και το σεβασμό μας για τη δουλειά που κάνατε και την αφοσίωση που δείξατε υπέρ της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε για λίγο και θα συνεχίσουμε μετά με τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. just... Παρακαλώ, καθίστε συνάδελφοι για να αρχίσω με την ψηφοφορία. So, ich darf Ihnen vorab mitteilen, να σας ανακοινώσω καταρχήν ότι οι Επιτροπές ΕΚΟΝ και ΕΝΒΙ αποφάσισαν πριν από την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο να αρχίσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις ε, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού. Η θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, που είναι και η εντολή για τις, διαπραγμα... τις διαπραγματεύσεις αυτές, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος του θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Ε, έκθεση Μπλίνκεβιτσιούτε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Is this no? Can I close? Πέρας της Δεκτή. Περνούμε στην επόμενη έκθεση του συναδέλφου Ντέιβις για το δίκαιο της αλληλείας, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τα αλληλευτικά δικαιώματα. Ich schließe die... της ψηφοφορίας. δεκτή και αυτή. Προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Βαν Όβερτφέλτε για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης το 2020. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Και αυτή η έκθεση έγινε δεκτή και περνούμε στην ολοκλήρωση των ψηφοφοριών κατεπήγοντος μετά από αίτημα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας δεκτή. Ευχαριστώ θερμά. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα. Σα ευχαριστώ. μικρόφωνο.